Colleagues, um, if you don't mind, I'm going to make a... αν δεν έχετε αντίρρηση, να αρχίσουμε, λέει ο Πρόεδρος. Να αρχίσουμε στην ώρα μας. Γιατί θα πρέπει οι προσκεκλημένοι μας να αποχωρήσουν και πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση να αρχίσουμε στην ώρα μας για τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ εσάς που ήρθατε στην ώρα σας, λέει ο Πρόεδρος. Το σημερινό θέμα είναι η στατική ιστορική ασφάλεια. Αρχίζουμε ευθύ αμέσω με αυτό το πρώτο θέμα μα, που είναι δραστηριότητε τη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακή συνεργασία. Θέματα ιστορική ασφάλεια. Η επιβολή του νόμου και εσωτερική ασφάλεια. Έχουμε την εισήγηση που θα κάνει ο κύριος Πιαντεντόζη, ο οποίος είναι ο προεδρεύων ε, λόγω Ιταλικής Προεδρίας και επίσης έχουμε και τον κύριο Ράιτ που είναι ο διευθυντής της Europol. Όπως γνωρίζετε συνάδελφε, η εσωτερική ασφάλεια είναι το θέμα το οποίο είναι πολύ ψηλά ε, όσον αφορά το πολιτικό μας θεματολόγιο, τις προτεραιότητές μας και ξέρετε είχε γίνει αρχή συζήτηση πριν από την προφορική ερώτηση. Οπότε και έτσι νομίζω θα έχουμε μπροστά μας όλο το φάσμα των μέτρων που χρειάζονται για την πλευρά της την επιχειρησιακή. Είναι εδώ λοιπόν εξ ο κ. Πιαντεντόζη, ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής, που, Κόζη, που συγκροτήθηκε δύναμη του άρθρου 71 της ε, συνθήκης συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο τόσο να εξασφαλίσει ότι θα αναβαθμιστεί η συνεργασία σε αυτά τα ζητήματα και σας συμμεθυμίζω συνάδελφοι ότι αυτό έγινε για να διευκολύνει και να συντονίσει τη δράση των μικρών μελών και των αρμοδίων υπηρεσιών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρόκειται να μας κρατούν ενήμερους για τις εξελίξεις. Πρώτος θα λάβει το λόγιο στη συνέχεια ο κύριος Ράιτ, που πρόκειται να μας κάνει μια παρουσίαση, ε, συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρησιακής συνεργασίας, συγκεκριμένα δηλαδή για την επιχείρηση Αρχιμίδης που είναι αρκετά πρόσφατη και είναι η μεγαλύτερη συντονισμένη ε, επιχείρηση που έχει αναλυφθεί κατά το οργανωμένο εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από χίλιες συλλήψεις οι οποίες ε, ακολούθησαν από αυτή την ε, μία ε, επιχειρησιακή ενέργεια. Κύριε Πιαντιντόζη, έχετε τη σκητάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή την ακρόαση σε αυτό τον ε, χώρο. Οι προσέσεις έχουν γίνει ήδη, οι συστάσεις ε, είναι ο αρμόδιος ε, για τη δημοσία ασφάλεια στο Υπουργείο Ιστορικών με το ρόλο του συντονιστή των αστυνομικών δυνάμεων της Ιταλίας. Σήμερα όμως σας μιλάω ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την Επιτροπή σας που μου έκανε την τιμή να παρουσιάσω σε αυτή τη συνάντηση τα άλλα 27 μέλη της Επιτροπής, εκ μέρους των οποίων σας χαιρετώ. Όπως ήδη ανέφερε ο Πρόεδρος στην παρουσίαση, η ΚΟΖΗ ιδρύθηκε το 2010 μετά από τη θέση ισχύ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως καθήκον τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και οργανισμών της Ένωσης. Είναι μια επιτροπή σχετικά νέα, επιχειρησιακή, με εντολή που προβλέπεται από το άρθρο 71 της Συνθήκης για τη Λειτουργία και από την απόφαση του Συμβουλίου 131 του 2010. Η Επιτροπή επιπλέον διαθέτει μια δυναμική συνιστόσα και προσαρμόζει το θεματολογιό τη στις διαρκείς εξελίξεις των απειλών προς την εσωτερική ασφάλεια. Στην κόζη συναντώνται ε, ψηλόβαθμα στελέχη που ασχολούνται με την εσωτερική ασφάλεια για να εντοπίσουν τις κυρίες ε, απειλές προς την εσωτερική ασφάλεια και να μελετήσουν τους τρόπους αντιμετώπισης μέσω του μέσου πώληση cycle για το οποίο θα συζητήσουμε αργότερα με τον διευθυντή της Europol. Συναντώνται επίση ε, για να διευκολύνουν την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων οργανισμών της Ένωσης που ασχολούνται σε διαφόρου βαθμού με την εσωτερική ασφάλεια. Επίση, συναντώνται για να ενισχύσουν τι συνδέσμου μεταξύ τη εξωτερική και τη εσωτερική διάσταση ε, τη ασφάλεια ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να παράσχουν αξιολογήσει στο Συμβούλιο σε θέματα εσωτερική ασφάλεια. Από την ίδρυσή τη, από την ίδρυση της Επιτροπής συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους οργανισμούς ώστε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς σχεδιασμού, συντονισμού και εκτέλεσης ε, επιχειρηματικών δράσεων στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των σοβαρότερων απειλών προς την εσωτερική ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο ενοποιούμε και συντονίζουμε τις αποκρίσεις των επιμέρους κρατών μελών με τις αποκρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο της συνθήκης που ιδρύει την ΚΟΖΗ προβλέπει να αναφέρει τις δραστηριότητε της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρόσφατα εγκρινάμε την τρίτη έκθεση που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου του 2013 με Ιούνιο του 2014 και καλύπτει στην Ιρλανδική, Λιθωνική και Ελληνική Προεδρία. Συνοπτικά Βασίζεται η δραστηριότητά μας στη συνεργασία μεταξύ των διαφορών οργανισμών και των εθνικών αρχών. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το policy cycle που ανέφερα προηγουμένως, ένα σχέδιο πολιετές, συντονισμένο, πολυτομεακό, με στρατηγικές προτεραιότητες που ορίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών. Μετά από την πρώτη περίοδο ρονταρίσματος, τώρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις της τετραετούς περίοδου 2014-2017. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η επιχείρηση Αρχιμίδης, μια άνευ προηγουμένη επιχείρηση στην αντιμετώπιση, στη συντονισμένη αντιμετώπιση των σοβαρών, του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη, την οποία θα σας προσφέρει αργότερα ο κύριος Βέινραιτ. Δεν θα σας μιλήσω για το policy cycle και τις πτυχές που ήδη υπάρχουν στην έκθεση προς το Κοινοβούλιο. Αντιθέτως θα προσπαθήσω να σταθώ σε ορισμένα νέα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το τρέχον εξάμεινο Προεδρίας. Όπως ήδη είπα, ένα από τα χαρακτηριστικά της κόζη είναι η επιχειρησιακή της δραστηριότητα. η ικανότητά της ε, να προσαρμόζει την ατζέντα της της εργασίας της στις νέες προκλήσεις ασφάλειας και να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτές τις ε, απειλές. Γι' αυτό το λόγο τον περασμένο Ιούνιο το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε ένα έγγραφο για το μέλλον της ΚΟΖΗ όπου η Επιτροπή προσδιορίσε τις σημαντικότερες απειλές και τους τρόπους αντιμετώπισης των μεταξύ των σημαντικών αυτών ζητημάτων προσδιορίστηκαν, διακρίνουμε την τρομοκρατία πρώτα απ' όλα, για αυτό το κοινωνικό αλλά και εγκληματικό φαινόμενο η ΚΟΖ έχει τη δυνατότητα να παρέμβει με την υποστήριξη προς τις ομάδες του Συμβουλίου για συγκεκριμένα ζητήματα όπως οι ξένοι μαχητές, παρέχοντας πολυτομιακή στήριξη. Για παράδειγμα, διευκολύνοντα το συντονισμό τη απόκριση των διαφόρων ενδιαφερομένων για την αντιμετώπιση του ζητήματο της ριζοσπαστικοποίηση, την εξέταση των κοινωνικών πτυχών και ενισχύοντας ε, του συνδέσμους μεταξύ των ε, φορέων ασφάλειας και άμυνας. Επίσης ε, ασχολείται με το συντονισμό των διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια και που συνομιλούν με διάφορους ενδιαφερόμενους εντός των ενωσιακών δομών και μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ τους. Η ΚΟΖΗ ασχολείται με την παρακολούθηση αυτής της συνεργασίας ελέγχοντας κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών. Όλο αυτό φυσικά δυνάμει του ισχύοντος νομικού πλαισίου σε θέματα προστασίας δεδομένων. Ένα άλλο θέμα είναι η συνεργασία μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Πρόκειται για μια θεμελιώδη πτυχή και πραγματική προτεραιότητα της Ιταλικής Προεδρίας. Η ασφαλεία της Ένωσης, κυρίως η εσωτερική, είναι μία και ενιαία. Είναι η ασφάλεια των πολιτών της, των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Σε οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική πολιτική της Ένωσης, όταν αναφερόμαστε στο θέμα της ασφάλειας, οι βασικές αρχές και οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν είναι οι ίδιοι. Παρότι λαμβάνουν διαφορετικές μορφές τις διάφορες δράσεις. Εκεί λοιπόν είναι σημαντική η σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή είναι αναπτύσσει πολιτικές ε, για την εξωτερική διάσταση, όπου η ασφάλεια διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, η πολιτική διεύρυνσης και γειτονίας. Είναι σημαντική επίσης η σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με την Πολιτική Επιτροπή Ασφαλείας όσον αφορά την, πολιτική, την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Η βασική αρχή που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι οι μεγαλύτερες απειλές προς την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννώνται και εξελίσσονται εξωτερικά σε περιοχές ε, εμπόλεμες ε, και από εκεί προέρχονται οι ροές ε, παράνομης διακίνησης και οι εγκληματικές ροές. Ας μην ξεχνάμε τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων ή τις ομάδες που εκμεταλλεύονται την παράνομη μετανάστευση. Οι προκρίσει λοιπόν είναι παγκόσμια σε αυτό τον παγκόσμιο κόσμο και απαιτούν παγκόσμια απάντηση, απόκριση. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντική η εσωτερική συνεργασία, δηλαδή συνοχή μεταξύ όλων των μέσων της Ένωσης και η συνεργασία με τρίτες χώρες. Ορισμένες συγκεκριμένες δράσεις που προωθούνται υπό την Προεδρία μας είναι πρώτα απ' όλα η συνεργασία με την Ιντερπολ παγκόσμιο πρωταγωνιστή στη διεθνή συνεργασία αστυνομικών δυνάμεων. Το Συμβούλιο Υπουργών του Οκτωβρίου ενέκρινε μια πρόταση της ΚΟΖΗ για να γίνει πιο αποτελεσματική η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων της Ίντερπολ στους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια έχουμε τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ πολιτικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οργανισμών όπως Ευρωπόλ και Frontex. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με τους ε, εκπροσώπους της ε, Πολιτικής Επιτροπής Ασφαλείας, ε, στην οποία θα συμμετέχω και γι' αυτό θα ζητήσω, θα ζητήσω συγγνώμη που θα αναχωρήσω. Η ενίσχυση του ρόλου της κόζης στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές που συμμετέχουν των χωρών που συμμετέχουν στην πολιτική διεύρυνση. Αυτή είναι μια άλλη πολύ συγκεκριμένη δράση. Χθες μόλις συζητήσαμε στην Επιτροπή τα αποτελέσματα του Progress Report της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Στις εκθέσεις της Επιτροπής επισημαίνονται ορισμένοι κρίσιμοι τομείς που αφορούν τη διεθνή συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων των χωρών αυτών προσπαθούμε να διαμορφώσουμε συνεργατικές μορφές, ε, μορφές συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κρίσιμα προβλήματα. Μια άλλη πτυχή είναι ο καθορισμός ιδανικών ε, τρόπων εργασίας η Είναι η, Επιτροπή, η ανώτατη Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τεχνικό επίπεδο πρέπει λοιπόν να διατηρήσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επιχειρησιακών δυνατοτήτων ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Γι' αυτό το λόγο στο πλαίσιο της Επιτροπής υπάρχει σταθερή εστίαση στις μεθόδους εργασίας που μπορούν να διασφαλίσουν ταχύες και αποτελεσματικές απαντήσεις. Η τελευταία πτυχή στην οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, αξιότιμα μέλη, είναι ο ρόλος της ΚΟΖΗ στην ε, διαμόρφωση της νέας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας. Όπως συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς στο Συμβούλιο Τζάι τον περασμένο Ιούνιο, η Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας θα πρέπει να αποτελεί όλο και περισσότερο ένα αξιόπιστο σημείο αναφορά του Συμβουλίου Υπουργών για όλα τα επιχειρησιακά ζητήματα που σχετίζονται με την εσωτερική ασφάλεια και με την αστυνομική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Γι' αυτό τον λόγο η ΚΟΖΗ κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας συντόνισε τις δραστηριότητες ε, στις διάφορες ομάδες και επιτροπές του Συμβουλίου ώστε να εκπονηθούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη νέα στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου είχε κάνει έκκληση για την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας νέας στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας βασισμένη στη συνεργασία Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Η συμμετοχή του Συμβουλίου περιλαμβάνεται σε ένα κείμενο συμπερασμάτων που χθε εγκρίθηκε από την ΚΟΖΗ και που θα περάσει από το Συμβούλιο των Υπουργών του Δεκεμβρίου. Η Ιταλική Προεδρία της ΚΟΖΗ που εκπώνησε το αρχικό σχέδιο των συμπερασμάτων και που μερίμνησε για τις διαπραγματεύσεις ε, εστιάστηκε σε συγκεκριμένες αρχές. Πρώτη, η ανάγκη ύπαρξης ενός πολιτικού εγγράφου σχετικά σύντομου στρατηγικής σημασίας που θα καταδεικνύει τις αρχές και τα οριζόντια ζητήματα, τα εγκάρσια ζητήματα υψηλής σπουδαιότητας. Προτείνει μια, προτείνει ένα κατάλογο εγκλημάτων αλλά και μέθοδο προσδιορισμού των διαφόρων εγκληματικών φαινομένων στα οποία θα πρέπει να εστιαστούμε. Άλλη βασική αρχή ήταν η δομή που προτάθηκε για τη νέα στρατηγική, η οποία έχει ως εξή. Πρώτα απ' όλα προσδιορισμός των απειλών και των προκλήσεων μέσω του policy cycle. Στη συνέχεια η υιοθέτηση μιας πολυτομιακής μεθοδολογίας ε, απόκρισης στα διάφορα φαινόμενα βασισμένη στην πρόληψη και στην πρόβλεψη των ίδιων των φαινομένων βάσει ανταλλαγής πληροφοριών, ε, χρήσης των νέων τεχνολογιών και βάσει της ανάπτυξης της συνεργασίας με τον τομέα της έρευνας. Αυτό είναι κάτι που θεωρούμε πολύ σημαντικό για το μέλλον. Συντονισμός των ερευνών και των διαδικασιών, με κεντρικό ρόλο στη Europol και στη Eurojust. Συντονισμό με άλλες στρατηγικές θαλάσσια, ναρκωτικών, εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, τρομοκρατίας. Τέλος, ενοποίηση και υλοποίηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου αντί για δημιουργία νέων νομοθετικών εργαλείων. Ένα άλλο στοιχείο της δομής που προτείνεται είναι ότι στη στρατηγική περιλαμβάνονται οι αρχές που προανέφερα σε σχέση με τη σχέση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Δόθηκε ιδιαίτερη επισήμανση, για παράδειγμα, στην συνεργασία και επιχειρησιακή συνεργασία με τις τρίτες χώρες και ειδικότερα με τις χώρες εκείνες από τις οποίες προέρχονται ή διέρχονται οι διάφορες απειλές προς την εσωτερική ασφάλεια. Αυτό ειδικότερα για τα μεταναστευτικά ζητήματα, αλλά όχι μόνο και υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα συνοχής μεταξύ όλων των ενωσιακών πολιτικών σε θέματα ασφάλειας. Επισημαίνεται πράγματι η αναγκαιότητα για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πρεσβείων των κρατών μελών, των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως για παράδειγμα οι αστυνομικές δυνάμεις. Τέλος, το έγγραφο έφεστα ιδιαίτερα την προσοχή στο ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός χώρου προστασίας των πολιτών μας και σεβασμού των δικαιωμάτων τους. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και με την κοινωνία των πολιτών ώστε να έχουμε κοινωνική συμμετοχή και συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο η Ιταλική Προεδρία πρότεινε μέγιστη υποστήριξη από τον οργανισμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα που για πρώτη φορά κλήθηκε να συμμετάσχει στις εργασίες της ΚΟΖΗ. Αυτό είναι απαραίτητο κατά την απόψή μα, ώστε να υπάρχει συνεχή εξισορρόπηση των διαφόρων πτυχών ασφάλεια και τήρηση των δικαιωμάτων. Θεωρούμε ότι οι σημερινές προκλήσεις ε, προς την ασφάλεια των πολιτών σχετίζονται με την τήρηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, που είναι και ο λόγος, ο βασικός για τον οποίο υπάρχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση Ελπίζω λοιπόν ότι οι δράσεις της Κόζη που παρουσίασα θα βρουν σύμφωνη την αξιότιμη επιτροπή σας και είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ακούγοντάς σας, καταλάβαμε ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιε παρουσιάσει σε τακτά διαστήματα από την Κόζη, γιατί έχει περάσει ένα χρόνο από το τότε τελευταία φορά στην Επιτροπή μα, που πρόκειται για α, κάτι επιχειρησιακό και χωρί να προδικάζω ότι θα πούνε οι συνάδελφοι και θα πει ο κύριο Βουίνραϊτ, αλλά είναι φανερό ότι όποτε έρχεστε εδώ να μα μιλήσετε, θα πρέπει να συζητήσουμε τα επιχειρησιακά ζητήματα και να επισυργόμαστε στις ε, λεπτομέρειες για αυτή τη βάση δεδομένων, για τις διακινήσεις κλπ. Αλλά όλα αυτά με την επιφύλαξη των όσων θα πούνε οι συνάδελφοι στη συνέχεια κατόπιν και της ε, ε του κ. Wainwright, ο οποίος τώρα θα κάνει τη δεύτερη ε, επιχειρησιακή παρουσίαση. μας πήγε αυτή επομένως την ε, επιχείρηση Αρχιμίδες, την μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση που έχει λάβει ποτέ χώρα. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Good morning, uh, uh Καλημέρα σας συνάδελφοι. Εδώ πρόκειται για μια σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης uh, Αρχιμίδης όπου θέλουμε να παρουσιάσουμε το πώς εφαρμόζεται η ενωσιακή πολιτική στην πράξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτή την επιχείρηση. Όπως ε, πολύ καλά γνωρίζετε, ε, τεχνικά είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί στη Europol, όπως αποδείχθηκε και από την ομιλία που επιχείρησε να κάνει ο υποφαινόμενος. Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα ε, σε κάποια θέματα προσπαθώντας να καλύψω αυτή την εντύπωση που δημιουργήθηκε από την αρχή της ομιλίας μου να σας πω τι μπορούμε να προσφέρουμε και επίσης να αναφερθώ στο ότι ο συντονισμός γίνεται από τα κεντρικά γραφεία στη Χάγη. Πριν ε, από μερικές εβδομάδες έγινε μάλιστα ο συντονισμός ε, και αναπτύξαμε 25.000 άντρες στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική ανάπτυξη δυνάμεων για την επιβολή του νόμου στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί συμμετείχαν σε συντονισμένες δράσεις ε, σε πάνω από 300 ε, επιχειρήσεις ε, σε 260 περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πόλεις, σε αεροδρόμια, σε σημεία διέλευση των συνόρων και σε άλλα σημεία. Και με βάση τις πληροφορίες μας, αν θέλετε, είναι η μόνη συντονισμένη ενέργεια κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν αποτελεί ορόσημο στις προσπάθειές μας του να αναπτύξουμε συντονισμένες δράσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η κοινωνία και οι πολίτες μας. Αυτές ε, είχαν αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στην Ευρώπη από ε, διάφορους που επιχείρησαν να μετακινήσουν παράνομα ναρκωτικά μέχρι και μετανάστες στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της επιχείρησης, διάρκεια 9 ημερών το Σεπτέμβρη, η Europol και το κέντρο συντονισμού της Europol ε, οργανώθηκε στα κεντρικά μας γραφεία για αυτή την πολύ προχωρημένη δράση. Ανταλλάξαμε 1500 αιτήματα για ανταλλαγή πληροφοριών και το τελικό αποτέλεσμα ή τα αποτελέσματα εξακολουθούν να προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε αυτή την επιχείρηση των 9 ημερών προέκυψε από τα αιτήματα για σύλληψη 1.400 ε, τότωσων ε, ε, υπόπτων, 600.000 ήταν οι τόνοι των υπόπτων ναρκωτικών, επίσης υπήρξε κατάσκηση περίπου 140.000 ε, παράνομων, παράνομο πληθυσμού. 200 θύματα της ε, παράνομης εμπορίας ανθρώπων, οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 100 ε, έμποροι παράνομης εμπορίας συνελήφθησαν και συνελήφθησαν επίσης περίπου και 20 αυτοκίνητα. Επίσης ε, υπήρξαν και πάρα πολλές άλλες χώρες που συνεργάστηκαν με την Europol, η Κολομβία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, το Ηνωμένε Πολιτή, η Σερβία, η Interpol και πολλοί άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαδρομάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επιχείρηση, κυρίως η Frontex αλλά και η Eurojustice. Ε, οι προτεραιότητες λοιπόν που αναφέρονται στον κατάλογο των επιχειρήσεων αναφέρθηκαν από τον πρόεδρο της Κόζη και θα ήθελα λοιπόν να τους συγχαρώ για όλους αυτούς τους υπαλλήλους επιβολής του νόμου που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και σε άλλες χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και που συνέβαλαν όλοι ε, σε αυτή την επιτυχημένη επιχείρηση. Επίσης ε, θα ήθελα να συγχαρώ και τους εκατοντάδες υπαλλήλους της Europol που διευκόλυναν όλη αυτή την δραστηριότητα και συνέβαλαν στην επιτυχία της επιχείρησης. Συνολικά λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία ε, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται αυτή. Αυτά αναφέρθηκαν και από τον προαλήσαντα. Όταν είχαν ε, σχεδιαστεί και εγκρίθηκαν οι νέες ρυθμίσεις υπό την Βελγική Προεδρία και προέκυψε η νέα κοινότητα επιβολή του νόμου υπό την καθοδήγηση της Κόζη, είχαμε λοιπόν δύο βασικές επιταγές. Το ένα ήταν ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στι αρμόδιε υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Ένωση. η κοινότητα τη επιβολή του νόμου να είναι πιο συμπαγή από ποτέ. Και το, η δεύτερη επιταγή ήταν η στρατηγική στόχη τη πολιτική να μεταφράζονται σε συγκεκριμένε επιχειρήσει. Αυτό λοιπόν δεν ήταν απλά ένα στρατηγικό έγγραφο, αλλά ήταν ένα τρόπο για να προκύψουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία κατ' ουσίαν διαφοροποιούν και τι δικέ μα δράσει για την ασφάλεια των πολιτών μα. Η επιχείρηση Αρχιμή ήταν ε, πρωτοφανής ε, όσον αφορά το σχεδιασμό και τα αποτελέσματά της βεβαίως ανταποκρίθηκαν στα αναμενόμενα. Δεν πρέπει να πούμε ότι βέβαια η επιχείρηση δεν αντιμετώπισε δυσκολίες, κάποια πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε προγραμματίσει και το βασικότερο όφελος από αυτή την επιχείρηση ήταν να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες της ε, κοινότητας επιβολής νόμου σε ένα πραγματικό σενάριο, ε, σε ένα ρεαλιστικό σενάριο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τόσες πολλές χώρες. Εξακολουθούμε να μαθαίνουμε πάρα πολλά για το τι σημαίνουν όλα αυτά, για το πώς πρέπει να προγραμματιστούν στο μέλλον. Η επιχείρηση όμως Αρχιμίδης αλλά και πολλές άλλες ε, διασυνοριακές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι τώρα αρχίζουν να αποδίδουν όλα αυτά και η κοινότητα της επιβολής του νόμου οριμάζει όσον αφορά τον συμπαγή της χαρακτήρα και τη γενικότερη αποτελεσματικότητά της. Νομίζω λοιπόν βράχει πρόθεσμα, προχωρήσαμε. Ο κύκλος πολιτικής εξακολουθεί να είναι μια πολιτική αλλά αρχίζει να λειτουργεί στην πράξη. Και επίσης πιστεύω ότι η Europol τώρα ε, γίνεται το κέντρο συντονισμού για πολλές ε, διεθνείς ε, επιχειρήσεις και για την επιβολή του νόμου στην Ευρώπη. Παράλληλα, ενώ υπάρχει η συμμετοχή και άλλων σημαντικών εταίρων, ε, βλέπουμε ότι συμμετέχουν κυρίως οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στη Χάγη σιγά σιγά ε, φτιάχνουμε ένα κέντρο για την Ευρώπη και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως με χαρά μας συμβάλλουμε σε αυτή την επιχείρηση και θέλουμε να συνεργαστούμε για την επιτυχημένη επιβολή της εφαρμογής του νόμου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βουέντρα, ευχαριστούμε που ήσασταν σύντομος. Τώρα λοιπόν μπορεί να προκύψει η ανταλλαγή απόψεων. Ας ξεκινήσουμε ε, καταρχήν με τον κύριο Κέκχοπ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα ε, να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές ε, για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που έκαναν και για την περιγραφή των θεμάτων. Σύντομες θα είναι οι παρατηρήσεις μου και ας επικεντρωθούμε σε κάποια θέματα που είπε ο κύριος Wainwright για τον Αρχιμίδη, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι θέλει να συνδυάσει αυτούς όλους τους οργανισμούς όπως μας περιέγραψε βεβαίω και θέλω περαιτέρω τώρα να μας πει και να μας περιγράψει τι γίνεται με την προσθεμένη αξία του να δουλεύουν όλοι αυτοί οι οργανισμοί σε συνεργασία γιατί έχοντας όλο αυτό το πλαίσιο πολλές φορές έχουμε τον κίνδυνο της έλλειψης του συντονισμού. Αυτό πώς το ξεπέρασε. Γιατί όλα αυτά τα επιδέματα, πάνω από χίλιες συλλήψεις, ε, τι γίνεται με τα ζητήματα για ναρκωτικά, για ελαθρομετανάστευση, όλα αυτά τα οποία ε, προέκυψαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα, ε, τόσα, τόσα, τόσα εγκλήματα τα οποία συνεχίζουν η Εθνική Αστυνομία ή η Europol σε ειδικέ περιπτώσει υπό την διοίκησή του. Οπότε θα ήθελαμε πάνω σε αυτό να μα πει τι γίνεται, γίνεται με την προσθέμενη αξία τη συνεργασία των αυτών των αρχών. Εντάξει, ε, ονομάζεται η επιχείρηση, αλλά εγώ θα ήθελα να μάθω κατά πόσο αυτό θα είναι πάγιο, κατά πόσο θα είναι μακρόπνο, διαρκές ως ε, ρύθμιση. Τι πιστεύει ο κύριος Γουένρα πιστεύει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις, συμφωνίες για να συνεχιστεί αυτή η υπόθεση. Σημειακά ή σε διάρκεια θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ευχαριστούμε Τίμωθη Λεπρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Κόζη. Άκουσα τα όσα είπατε για την ανάγκη για ύπαρξη μιας ολιστικής προσέγγισης και ενοποίησης της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεδομένων των απειλών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και λαμβάνοντας υπόψη και την προέλευση των εγκλημάτων. Άκουσα επίσης το πώς υποστηρίξατε αυτή τη νέα προσέγγιση στην αναθεώρηση της ε, στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και για τη συνεργασία που απαιτείται μεταξύ κρατών μελών. Ναι, πράγματι γνωρίζουμε και πρόσφατα μάλιστα είχαμε μια άλλη ακρόαση όπου αναφέρθηκε ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικές δυσκολίες ε, σε πλαίσιο συνεργασίας, ε, για παράδειγμα όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών, αλλά και σε επίπεδο θα έλεγα άλλων ε, βασικών εργαλείων ασφαλείας όπως οι αστυνομικές δυνάμεις, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και εγώ τώρα μιλάω για την κατάσταση στη δική μου τη χώρα, στην Πορτογαλία, γνωρίζοντας πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυναμικά ε, δραματικά τις δυνατότητες απόκρισης όλων αυτών των δυνάμεων και αυτό έχει και συνέπειες και στη διαλειτουργικότητά τους. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι τι κάνετε στην κόζη για να διασφαλίσετε, ξέρετε δίνετε τόσο μεγάλη προσοχή ε, στα ευρωπαϊκά όργανα ε, εξετάζουν διεξοδικά το πώς λειτουργούμε οικονομικά και δεν βλέπουμε να υπάρχει τόσο μεγάλη παρεμβατικότητα όσο για την οικονομία όταν εξετάζουμε τα ζητήματα ασφαλείας των πολιτών μας. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο σε απειλές που αναφέρατε εσείς, αναφέρομαι και σε άλλες απειλές που οφείλονται σε άλλε εξωτερικές κρίσεις και που επηρεάζουν τη δική μας ασφάλεια. Για παράδειγμα, οι πτήσεις ε, ρωσικών μαχητικών πάνω από την επικράτειά μας και πώ θέτουν σε κίνδυνο κρίσιμε υποδομέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, τη λειτουργία του εναέριου χώρου μας ε, και οτιδήποτε πράγματος κυκλοφορεί εκεί. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τον κύριο Βέινραιτ... Δεδομένων λοιπόν όλων αυτών των απειλών, των εγκληματικών απειλών στις οποίες αναφερθήκατε, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες από παράνομες δραστηριότητες, σε ποιο βαθμό αποτελεί μέσο για να αντιμετωπίσουμε και άλλες μορφές εγκληματικότητες. Κυρίως όταν αυτή η νομιμοποίηση διευκολύνεται από το τρελό μας σύστημα, από την κατακαιρματισμένη φορολογική μας πολιτική, το κατακαιρματισμένα φορολογικά συστήματά μας που επιτρέπουν να ανθεί η εγκληματικότητα ελεύθερα. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, μπορεί να απουσιάσω για 10 λεπτά, αλλά θα επανέλθω να σας ακούσω. Okay, thanks, Να σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ έχουν ε, ζητήσει το λόγο, αλλά πρέπει να κλείσουμε στις 10. Άλμπρεχτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις. Έχω μία ερώτηση για τον καθένα. Πρώτη ερώτηση. Για τον κύριο Εντεντούτη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Πιαντεντόζη. Πέστε μας. Τι ισχύει δύναμη της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, γιατί διαπιστώνουμε ότι τα περισσότερα σε σχέση με την αστυνομία και την δικαστική συνεργασία είναι αντικείμενο συναπόφαση από το Κοινοβούλιο. Για να δούμε και να παρακολουθήσουμε τι γίνεται για αυτά τα μέτρα. Πώς θα γίνεται καλύτερα η έγκριση και η υλοποίηση να δούμε πώς θα έχουμε μια συνεργασία αναβαθμισμένη, ισχυρή, συνεχή μεταξύ ημών και της κόζη. Βεβαίω, πολύ ευχαριστώ να τα συζητούμε που καθόμαστε τώρα εδώ. Αλλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερο, τόσο ώστε να μπορούμε να προγραμματίσουμε καλύτερα τι γίνεται με την δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Άρα θα πρέπει να προγύψουν κάποιε ε, Συγκεκριμένε προτάσεις για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τι εξέλιξεις. Τώρα, δεύτερο για τον κύριο Γουένραϊτ. Είμαι θαυμαστή των όσων κάνετε, κυρίω όσον αφορά το κέντρο κύβερνο εγκλήματο. Τόσε ιδέες μου ήρθαν ε, τώρα που συζητούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πιο απάντως θα ήθελα το εξής, να σας τονίσω. Από δική μου πλευράς, και νομίζω ότι πολλοί συμφωνούν, εσείς, κατά κάποιο τρόπο αμαυρώνετε σχέση της προσπάθειας ε, γιατί τους δίνετε λάθος όνομα. Να, μας ε, μοιράσατε αυτό εδώ το φυλάδιο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, τη σχετική στρατηγική και Διάβασα το περισσότερο από αυτό το έργο και μετά λέτε η κατάχρηση της ανωνυμίας. Γιάν, Γιάν, πρέπει να σου πω, λέει ο πρόεδρος, ότι αυτό θα συζητηθεί στις 10 και μισή. Και θα είναι εδώ ο κ. Γουίνραιτ. Α, ωραία, ωραία, λέει ο κ. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί συνέχεια να τσεκάρει την ενέργεια. διαδεκτά, αλλά τέλο πάντων για αυτό έχετε τον πρόεδρό σα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ μερικά από αυτά που είπατε, αλλά με καλύψατε και σα ευχαριστώ. Συνάδελφοι, τηρήστε το χρονικό όριο των δύο λεπτών, γιατί έχουμε πάρα πολλού ε, να λάβουν το λόγο. Βέβαια, όλοι λέτε πολύ αξιόλογα πράγματα. Βερζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους δύο μιλητές μας. Όλοι είμαστε πεπισμένοι εδώ ότι τα δικαιώματα στην, στην ασφάλεια είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Τα δικαιώματα όμως αυτά πρέπει να υλοποιούνται με τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Το δικαστήριο το έχει υπενθυμίσει όσον αφορά τις δυσανάλογες υποχρεώσεις για τις ε, δράσεις τηλεπικοινωνιών και παρατηρούμε ότι όλοι προσπαθούν να κάνουν ότι μπορούν καλύτερο και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. αυτό δεν θα γίνει μόνο μέσω της κατάρτισης των ε, ε, υπαλλήλων αλλά με το να λαμβάνονται υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους τις πτυχές πολιτικές. Η Ένωση Δυνάμεων λοιπόν είναι σημαντική αλλά δεν είναι επαρκής κυρίως όταν συνίσταται σε μια συνεδρίαση εδώ και εκεί. Το θέμα είναι πώς γίνεται συνεργασία για παράδειγμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο με εκθέσεις κάπως καθυστερημένες και όχι αρκετά τακτικές πιστεύω ότι πρέπει να έρχεστε να μας αναφέρεστε πιο συχνά, σε κάθε προεδρία για παράδειγμα. Επίσης για να είμαστε υποτελεσματικοί χρειαζόμαστε πραγματικές, σοβαρές, συγκεκριμένες αξιολογήσεις συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των απειλών. Δηλαδή πραγματική αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα κράτη-μέλη. Διαφορετικά συντονισμός δεν σημαίνει τίποτα. Επίσης ε, αναφερθήκατε σε συνεργασία των ενδιαφερομένων. Ποιων ενδιαφερομένων τακτικά ε, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, μας στέλνουν προειδοποίησεις για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω έχουμε παραπάρει φόρα για να αντιμετωπίσουμε σοβαρούς κινδύνους στους οποίους εστιάζουμε τα μέσα εις βάρος άλλων πολιτικών και η συνάδελφός μου Αναγκόμες το υπογράμμισε για την περίπτωση της Πορτογαλίας. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το θέμα και πώς οι εσωτερικές προτεραιότητες, τις οποίες δεν πρέπει να παραμελούμε, θα συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη, όχι όμως εις βάρος άλλων επιγόντων σοβαρών ζητημάτων, αλλά που συχνά ε, ε υλοποιούνται με δυσανάλογα μέσα. Ευχαριστούμε η κυρία Άνς Κορνίλια. Έχω τρεις ε, ερωτήσεις που συνδέονται μεταξύ τους. Μιλήσατε για την επιχείρηση Αρχιμίδης. Απευθύνομαι στον κύριο Wainwright. Η Europol εργάζεται, συνεργάζεται στενά με την Frontex, το είπατε κι εσείς, και μιλάμε για 10.000 ε, παράνομους μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν, ελέγχθηκαν. Ίσως μπορείτε να μας ενημερώσετε λιγάκι καλύτερα από αυτού. Πώς ακριβώς συνεργαστήκατε με τη Frontex και μπορείτε να μας ενημερώσετε και για τους ε, πάνω από χίλιους ε, έγκλειστους ε, τους οποίους ε, έχετε εσείς βάλει στη φυλακή. Πώς ακριβώς ε, συντίθεται το ποσοστό της εγκληματικότητας στους χίλιους, γιατί από τους χίλιους πόσοι είναι εγκληματίες. Και αυτό που με ενδιαφέρει επίσης είναι το κόστος της επιχείρησης. Δηλαδή μια τέτοια επιχείρηση πόσο ακριβώς κοστίζει και τι είδους κονδύλια χρησιμοποίησατε για να αναπτύξετε αυτή την επιχείρηση. Ευχαριστούμε την Κορνίλια επόμενος είναι ο κύριος Κάρλος. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριος Κοέλιο. Πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι τα ε, σχόλιά σας ε, σχετικά με την επιχείρηση Αρχιμίδης ως ε, ένα εργαλείο για να συντονιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις με τη Europol. Επίσης, ο διευθυντής της Europol ανέφερε ότι αυτό ήταν μια ευκαιρία για να δοκιμαστούν στην πράξη η αντίδρασή μας μεταξύ άλλων και ελπίζω η Europol να έμαθε από την εμπειρία της. Ε, δεν είμαστε και πολύ εντυπωσιασμένοι από τα αποτελέσματα. 25.000 αστυνομικοί συνέλαβαν πάνω από χίλιους ανθρώπους, αλλά για να είμαι ειλικρινής, το περίπου 30% εξ αυτών είναι απλά λαθρομετανάστες, δεν είναι πραγματικοί εγκληματίες. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, όπως θα μπορούσαν να είναι, η σημασία αυτής της εμπειρίας έγκυται στο ότι πρόκειται για την πρώτη τέτοια κλίμακα επιχείρηση. Και η ερώτησή μου προς τον διευθυντή της Europol είναι η εξής. Ε, πρόκειται η Europol να καταθέσει μία έκθεση αναλύοντας τι πήγε καλά και τι όχι. Επίσης θέλω να ρωτήσω κατά πόσον την την έκθεση, θα τη δούμε και εμείς ή μήπως ε, θα έχει πρόσβαση αυτές τις πληροφορίες μόνο το Συμβούλιο. Πολύ. Ευχαριστώ κύριε ε, Κοέλιο. Θα ήθελα να συμφωνήσω λιγάκι με τους προλαλήσαντες με την έννοια ότι η επιχείρηση Αρχιμίδης είναι μια αστυνομική επιχείρηση με την οποία υποτίθεται ότι εντοπίζονται εγκληματίες. Βλέποντας όμως ότι μιλάμε για πάνω από χίλιους ή μάλλον χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι συνελήφθησαν, αλλά μόνο οι χίλιοι εξ αυτών εγκλίστηκαν στις φυλακές, υπάρχει εδώ μία δυσαναλογία. Και δεν θέλω τώρα να ρωτήσω τι έγινε τελικά με αυτούς τους υπόλοιπους μετανάστες, τους 9 περίπου χιλιάδες ε, οι οποίοι δεν προέβησαν σε αξιόπινες πράξεις. Ούτε καν θέλω να ρωτήσω. Όμως αυτή η χίλιοι, οι έγκλειστοι, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ για να ξέρω κατά πόσο δικαιολογείται όλη αυτή η δαπάνη. Δηλαδή, δεν θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες μόνο για ποια πράξη καταδικάζονται ή κατηγορούνται, αλλά θέλω να ξέρω κατά πόσον αυτοί ήταν οι εγκέφαλοι ή απλά τα εκτελεστικά όργανα, γιατί είναι δυνατόν και οι χίλιοι εξ αυτών να είναι πραγματικά ύποπτοι, να ξεκινήσει η κανονική δικαστική διαδικασία εναντίον των και πράγματι να καταδικαστούν τελικά για μια αξιόπινη πράξη. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και του άλλους ανθρώπους που επιτήρουν το, χρονικό όριο. Και τώρα ο κύριος Ντεπρέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όσον αφορά αυτούς τους κυβερνοεγκληματίες ε, ή να το συζητήσουμε με το επόμενο θέμα της μέσης διάταξης. Κύριε Πρόεδρε. Στις 10.30, 10.30 λέει ο Πρόεδρος. Για αυτούς τους κυβερνοεγκληματίες. Γι' αυτό το θέμα να το ρωτήσω για το επόμενο. Στις 10.30 δύο λέει ο πρόεδρος, στις 10.30. Μάρτζι Λόρεστον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την καινούργια κατάσταση, τις ευκαιρίες. Εγώ κάτι θέλω να ρωτήσω όσον αφορά την ασφάλεια, κάτι το οποίο έχει την εξωτερική και εσωτερική πτυχή όπως αναφέρατε στην παρουσίασή σας για την κόζη. Είναι και το θέμα της ψυχολογικής άμυνας, ψυχολογικής ασφάλειας. Υπάρχει κάποιος οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λαμβάνει υπόψη κάποια ζητήματα όπως σαν τον πόλεμο της πληροφορίας που γίνεται τώρα από διάφορες χώρες όπως χθες ας πούμε η Ρωσία ανοιχτά παρουσίασε μια στρατηγική ιντερνετική και διαφήμισε την καινούργια εποχή όσον αφορά ε, μέσω του Ιντερνετ δηλαδή θα παρουσιάσει τη, χώρα, ε, τη Ρωσία δηλαδή θα παρουσιάσουν οι Ρώσοι σε 45 χώρες και αυτό φυσικά πρόκειται να έχει επιρροή σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για μια προπαγάνδα που χρησιμοποιούν τώρα και στην Ουκρανία και άλλο. Υπάρχει κάποιος οργανισμός που ασχολείται με τον πόλεμο της πληροφορίας και την ψυχολογική άμυνα. Μάρτζη, σε ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Τόμισιτς, είστε ο επόμενος. Um, Ευχαριστώ πολύ. Όλες οι χώρες έχουν κάποιο είδου μαφία, αλλά σε ορισμένες ειδικότερα στις πρώην χώρες ε, λέμε ότι κάθε μαφία έχει μια χώρα. Γνωρίζοντας αυτό, ήθελα να μου πείτε, όταν γνωρίζετε ότι σε ορισμένες χώρες οι μαφίες συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις, πώς κάνετε την έρευνα όταν πηγαίνετε στη χώρα. Οι αξιωματήχοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ιντερπολ ή η Ευρωπόλ βρίσκεται εκεί ή πηγαίνετε incognito. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συναδέλφοι. Απλά να ελέγξω κατά πόσο μίλησαν όλοι όσοι ζήτησαν τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πειθαρχία σας και που τηρήσατε τους χρόνους. Έχουν μιλήσει όλοι. Έχουμε και άλλα σημεία. Έχουμε μια προφορική ερώτηση και ένα σημείο στην ημερησία διάταξη για το έγκλημα στον χώρο. Οπότε και εκεί θα επανέλθουμε στο ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας. Εγώ ήθελα να πω ότι είναι σαφές από τις ερωτήσεις που ακούσαμε ότι επανέρχονται κάποια ζητήματα. Υπάρχουν νέα μέσα της Επιτροπής για τη διακίνηση ανθρώπων, δεν έχουμε εξετάσει το ζήτημα των ξένων μαχητών, τι έχει γίνει στο Συμβούλιο, στην Κόζη, για το ζήτημα αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει τους συναδέλφους. Κύριε Διάσταμαρη, θέλατε να πείτε κάτι γι' αυτό τώρα. Παρακαλώ, γρήγορα. Δίας ε, Σύντομα κύριε Πρόεδρε, όχι εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ για το Αρχιμίδης. Απλώς θα ήθελα να σας εκφράσω την περίεργειά μου. Θέλω δηλαδή να μάθω ποια θα είναι η αποτελεσματικότητα του έτσι Όπου θέλω να ρωτήσω τον διευθυντή του Κόζη, γιατί ακούσαμε ότι θα πρόκειται για ένα σύντομο, στρατηγικό, οριζόντιο έγγραφο. Ε, και εκεί θα έχουμε ένα κατάλογο εγκλημάτων ε, και άλλα. Θα περιέχει ειλικρινά. Θεωρώ ότι υπό τη σημερινή συγκυρία, στο σημείο που βρισκόμαστε, είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Να δούμε Εάν το Δεκέμβριο πρόκειται να χτυπήσει το καμπανάκι στο Συμβούλιο με αυτό το έγγραφο και η ΛΥΜΠΕ επίσης να δει ακριβώς ε, αυτό το έγγραφο πόσο ενδελεχές είναι και να δούμε τι γίνεται με κάποια βασικά ζητήματα που έχουν βέβαια σχέση με την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ και το τελευταίο που θέλω να πω είναι αυτό που ο κύριος Άλμπρεκτς ε, αναφέρθηκε στο ότι Πώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνομοθέτη μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα με το Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι όταν επανέλθουμε μπορούμε να κοιτάξουμε πιο πολύ σε βάθος ορισμένα από αυτά τα σημεία. Έχετε το λόγο κύριε Πιάντεντόζη και μετά θα ζητήσουμε από τον κύριο Wainwright να απαντήσει κάποιε από τι ερωτήσει. επίση. Θα περιοριστώ σε μια συνοπτική απάντηση προσπαθώντας να απαντήσω φυσικά τα πάντα αλλά θα προσπαθήσω φυσικά να απαντήσω όσο γίνεται πιο διεξοδικά το ευρύ φάσμα των ερωτήσεων των ε, βουλευτών εδώ. Πολλές από αυτές τις ερωτήσεις διασυνδέονται μεταξύ τους. Θα εμπνευστώ και από τα μέσα πληροφορικής που έχουμε επίσης ε, εγώ έχω να πω ως πρόεδρος της ΚΟΖΗ θα είμαι στη διάθεσή σας και αργότερα για να σας στείλω και γραπτές απαντήσεις ώστε να απαντήσουμε διεξοδικά όλες τις ερωτήσεις σχέση με τα όσα είπαμε σήμερα και φυσικά θα έχουμε και μελλοντικά ραντεβού στο πλαίσιο των σχέσεων μας με το Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στο τελευταίο σημείο της ε, παρουσίασής σας, η κόζη, όσον αφορά τους μηχανισμούς συναπόφασης η ΚΟΖΗ έχει επιχειρησιακό ρόλο. Δεν ασχολείται με με ε, βάση της συνθήκης δεν ασχολείται με νομοθετήματα ούτε συμμετέχει στη συναπόφαση. Η ΚΟΖΗ ασχολείται λοιπόν όχι με νομοθετικά θέματα αλλά με επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, οργανισμών και αρχών των κρατών μελών. Οι σχέσεις με το Κοινοβούλιο ρυθμίζονται λεπτομερώς από πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει το Συμβουλίο Υπουργών. Αλλά όπως είπα είμαστε διατεθειμένοι για ενημέρωση βάσει του σημερινού συστήματος ε, και βάσει των περιοδικών εκθέσεων. Είμαστε λοιπόν απόλυτα στη διαθεσή σας. Βάσει των μηχανισμών και των δομών που προβλέπει η συνθήκη και βάσει των αποφάσεων του Συμβουλίου, τις οποίες εμείς πρέπει να σεβόμαστε. Η Πορτογαλίδα βουλευτής ε, αναφέρθηκε στις δυσκολίες, τις οικονομικές δυσκολίες ε, των αστυνομικών αρχών λόγω της κρίσης αναφέρθηκε στο γεγονό ότι τα ευρωπαϊκά όργανα παρεμβαίνουν περισσότερο για τα οικονομικά θέματα και λιγότερο για τα θέματα ασφαλεία. Ήθελα να επισημάνω λίγο την ιδιαιτερότητα των μηχανισμών ε, αποτελεσματικότητας των αστυνομικών δυνάμεων. Εμείς γνωρίζουμε όλα τα αρνητικά πόσα εγκλήματα γίνονται στο πλαίσιο επιχειρήσεων όπως αυτή που ανέφερε ο Ρόμπ, η επιχείρηση Αρχιμίδης έχουμε και εκεί τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορούμε να συντονιστούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Αλλά κανείς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναφέρει με πλήρες λεπτομέρειες τι ακριβώς επέτυχαν οι δράσεις της, ε, των δυναμιών της τάξης. Ας δούμε την τρομοκρατία. Ένα τρέχον θέμα. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται την απειλή Φυσικά όταν συμβαίνει κάτι ανησυχητικό, κάτι ορατό, αλλά πολύ συχνά είναι αδύνατο να αναφέρουμε οτιδήποτε επιτυγχάνεται μέσω των δράσεων αυτών. Εγώ αναφέρω τον ε, τρομοκρατία, όχι γιατί είναι κάτι επίκυρο, αλλά γιατί εξορισμού χρειάζεται κάποια διακριτικότητα σε αυτές τις διαδικασίες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Ε, οπότε χρειάζεται κάποιος συντενισμός ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκεί αντιμετωπίζουμε εμείς ένα διπλό πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμούς, να τροφοδοτήσουμε μηχανισμούς ε, καθησυχασμού των πολιτών μας και να μην δίνουμε και τη λανθασμένη ιδέα ότι έχουμε θεσμικά όργανα ή εθνικές αρχές που σήμερα δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Δεν συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να βρισκόμαστε στο ύψος της απειλής που υπάρχει. Πρέπει να προσπαθούμε να προβλέψουμε τις πράξεις τρομοκρατίας. Εμείς κάνουμε σημαντικό έργο, επίσης σε μια πρόσφατη απόφαση του τελευταίου Συμβουλίου Υπουργό στο σημείο 13 του Roadmap που χαράχθηκε στο Συμβούλιο Τζάι τον Οκτώβριο. Εκεί τα κράτη-μέλη αποφάσισαν να δώσουν εντολή στην Προεδρία να διερευνήσει τις δυνατότητες διαφυλάσσοντας τη λειτουργικότητα των μέσων και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που σήμερα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες στα κράτη-μέλη, τη δυνατότητα λοιπόν δημιουργίας στην Ευρωπόλ μιας κοινή πλατφόρμας και για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Να σας αναφέρω μια δήλωση ενός συναδέλφου. ξέρω ότι στους μη ειδικού αυτά μπορεί να είναι λίγο δυσνόητα. Εμείς προσπαθούμε να εξορροπήσουμε τα πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε οι κύριοι φορεί να είναι τα κράτη-μέλη με τις υπηρεσίες πληροφοριών τους και τις υπηρεσίες της τάξης τους αλλά το πεδίο το δημιουργεί η Ευρωπόλ ε, το γήπεδο το δημιουργεί Ευρωπόλο ώστε να μπορέσουν να παίξουν καλύτερα εκεί οι διάφοροι παίκτες, οι διάφορες δυνάμεις ε, οι αστυνομικέ δυνάμεις της κάθε χώρας. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Διότι οι δομές, οι εθνικές νομοθεσίες, οι εθνικές αρχές ε, έχουν πολλές μορφές. Δεν είναι αρνητική η πολυμορφία πάντα στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, εδώ και δεκαετίες υπάρχουν θεσμικά όργανα που ασχολούνται με όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν παραδόσεις, κάποια κληρονομιά και εμπειρίε. Δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε αυτά. Γι' αυτό είναι σημαντικό συντονισμό που μερικέ φορέ ακούγεται κάπω ασαφή, όχι πολύ κατανοητό, αλλά αυτό είναι το στίχημα που πρέπει να παίξουμε. Πρόσφατα αναφέρθηκε, έχουμε, έχουμε πια στο θεματολογιό μας ότι οι διάφοροι φορείς, τα κράτη-μέλη πρέπει να βάλουν από κοινού τους σπόρους έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί η αποτελεσματικότητα των δυνάμεων επιβολής του νόμου λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο συντονισμός είναι αναγκαίος γιατί πρέπει να είναι πολυτομεακός. Γιατί ορισμένοι από εσάς ανέφεραν τα προβλήματα της διεύρυνσης, για παράδειγμα. Τα προβλήματα της διεύρυνσης είναι και προβλήματα ασφάλειας. Ασχολείται με αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι χρηματοδοτεί προγράμματα μέσω των οποίων τα κράτη-μέλη που προσπαθούν να βελτιώσουν τις ε, ικανότητες, τις διάφορες δεξιότητες και ικανότητες των κρατών ε, που συμμετέχουν στη διεύρυνση, το χρησιμοποιούν αυτό για να ελέγξουν και την ετοιμότητά τους, την επάρκειά τους ε, σε θέματα διεύρυνσης. Όπως βλέπετε όλα αυτά τα θέματα λοιπόν είναι αλληλένδετα. Και εκεί οι θέματα ασφαλείας και που αφορούν και την σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών είναι σημαντικά θέματα που ανατίθενται στις δυνάμεις της τάξης είναι θέματα που ξεπερνούν τα όρια της εσωτερικής ασφάλειας. Αυτή η διατομεακότητα, αυτός ο διατομεακός χαρακτήρας και συγγνώμη που απαντώ με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το θέμα λοιπόν ε, του εγκάρισου χαρακτήρα όλων αυτών των δράσεων αφορά τις σχέσεις μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Είναι σαφές ότι μπορούμε να αναλύσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι ανέλησα εγώ το γεγονός ότι σήμερα τα προβλήματα εσωτερικής ασφάλειας προέρχονται από περιοχές εξωτερικές. Οι ξένοι μαχητές είναι πρόβλημα τέτοιου είδους. Γνωρίζουμε όλοι ότι πρόκειται για δεύτερη γενιά ή τρίτη γενιά Ευρωπαίοι πολίτες όμως που πηγαίνουν να πολεμήσουν σε άλλες χώρες και μετά να γυρίσουν. Αποτελούν ένα πρόβλημα ασφάλειας που προέρχεται εκτός των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά που δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σοβαρά στις δικές μας χώρες. Είναι σημαντικό ζήτημα. Τώρα σας ζητώ συγγνώμη βέβαια γιατί θα πρέπει να λείψω για λίγο γιατί στις 10 έχουμε μια συνεδρίαση κοζικόψη δύο οργανισμοί της Ένωσης που ασχολούνται με την εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια και εκεί θα συζητήσουμε για το πώς θα βελτιώσουμε τις αποστολές ε, της αστυνομίας στο εξωτερικό. Δηλαδή το πώς μπορεί να συμβάλλει το σύστημα ασφάλειας για τον καθορισμό των αποστολών που θα γίνονται σε αυτές τις χώρες. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της συνεργασίας με τις ε, τρίτες χώρες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ε, τα προβλήματα της μετανάστευσης είναι προβλήματα ασφάλειας. Ε, νομίζω στην Ιταλία έχουν όλοι στραμμένοι το βλέμμα, γιατί η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει σύνορα στη Μεσόγεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενημερωθεί για το πρόβλημα αυτό. Το γνωρίζει. Γνωρίζει λοιπόν ότι με ένα και μόνο ε, φαινόμενο, το φαινόμενο της μεταφράστευσης. Προκύπτουν και πολλά άλλα προβλήματα. Είναι το θέμα του πώς υποδέχεται κανείς αυτούς τους μετανάστες, ε, πώς τους ε, εντάσσει και άρα δηλαδή πώς ρυθμίζεται και η σχέση με τις τρίτες χώρες. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, επίσης έγινε αναφορά στην στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια. Η δουλειά που γίνεται σε επίπεδο κόζη είναι η προετοιμασία ενός εγγράφου που θα έχει ουσιαστική πολιτική και στρατηγική σημασία. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, Συμβούλιο Υπουργών, άρα δηλαδή έχει μεγάλη, μεγάλο πολιτικό βάρος, πρέπει να προετοιμάσει τα συμπεράσματα της στρατηγικής και να μην είναι μια στρατηγική η οποία θα περιορίζεται μόνο στις ε, συνεισφορές όλων αλλά και σε αυτήν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σας είπα ότι μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό οικοδόμημα και αυτό απελαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η στρατηγική παρουσιάστηκε σε μια σύντομη συνάντηση που είχαμε. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πολιτικό έγγραφο άρα δηλαδή θα πρέπει να έχει και κάτι το πρωτότυπο, το μοναδικό, ένα σημείο κίνησης από το οποίο θα ξεκινήσουν όλες οι επόμενες δράσεις και το θέμα το οικονομικό. Όλα τα κονδύλια που θα πρέπει να διατεθούν και ένα μεταξύ άλλων παραδείγμα ήταν η επιχείρηση ε, Αρχιμίδης. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική της εσωτερικής ασφάλειας, εδώ πρόκειται για το θέμα κυρίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξέρετε, δεν είναι ότι δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Έχετε κάποιο διαδικαστικό, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Ντία Ντεμέρα, ναι σας ευχαριστώ. Ναι, είναι σχετικό με αυτό το σημείο. Κοιτάξτε κύριε Διευθυντά, εγώ μίλησα για το ΕΣΥ. Mm -hmm. Γιατί ακριβώ σεβόμαστε αυτό το οποίο πρέπει να αποχωρήσετε. Και πρόκειται για το επόμενο σημείο στη διάταξη. Πάντω είναι για μα πάρα πολύ σημαντικό να δούμε για την στρατηγική ιστορική ασφάλεια πώς θα διαμορφώσουμε αυτή μας την προφορική ερώτηση γιατί ε, πρόκειται να ακολουθήσει σοβαρή συζήτηση από αυτού και αυτό το οποίο εσείς είπατε ε, για την ε, στατική για όλα αυτά που μας αναφέρατε για ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα όπου προχωρήσατε μετά για μένα αυτό μου φαίνεται στοιχειώδες, στοιχειώδες σας το λέω με όλο το θάρρος και ε, μας, αυτό μας καίει. Και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και την προφορική ερώτηση, γιατί γι' αυτό και εγώ άλλωστε ε, κατά κάποιο τρόπο ε, προέτρεξα το προηγούμενο σημείο γιατί ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο το, το κοινοβούλιο τον ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπατε κύριε Ντίες και πριν ολοκληρώσετε ε, κύριε Σιγητά, ε, βλέπω ότι πολλούς βουλευτές απασχολεί το εξής. Ε, είχαμε μία παρουσίαση της Ξέρω πολύ καλό ότι πρέπει να φύγετε. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. θέλω όμως να πω ότι εδώ σήμερα μας κάνατε μία πολύ γενικευμένη, έτσι, γενικής φύσης παρουσίαση. Εδώ όμως πρόκειται για κάτι πιο συγκεκριμένο όπως αναφέρθηκε. Άρα δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουμε, τουλάχιστον όσο μας αφορά και οι ερωτήσεις γίνονται από τα μέλη μας, Όλα αυτά βασίζονται στο εξή. Εμεί θέλουμε να ξέρουμε τι θα κάνει το Συμβούλιο για την εμπορία ανθρώπων. Πρέπει να μπούμε σε βάθος σε αυτό το θέμα. Να διαπιστώσουμε ε, τι ακριβώς ε, γίνεται. Όχι να ενημερωθούμε για το α ή το β άρθρο να γίνει ουσιαστικό διάλογο. και ο κύριο Τεμέρα πολύ σωστά είπε ότι η στρατηγική εσωτερική ασφάλεια είναι μία από τι ε, μεγάλες μας προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν ε, θεωρώ ε, και από την έκφραση των προσώπων των συναντέλφων μπορώ να συμπεράνω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος επί του θέματος. Ίσως μπορούμε να κλείσουμε αυτή την παρατήρηση. Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς να προσθέσετε κάτι. Πάντως σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Δηλαδή ε, θα πρέπει ταχύτατα να επανέλθει εδώ η Κόζη, εκπρόσωποι της Κόζη. Παρακαλώ, εν πάση αν θέλετε κάποιες τελικές παρατηρήσεις, έχετε δυνατότητα να τις κάνετε. Κοιτάξτε, να είμαι ειλικρινής, ε, πιστεύω ότι κάποιες από τις ανησυχίες σας βασίζονται στην αναγκαιότητα να οριστεί σωστά ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την κόζη, αλλά κυρίως σε ποιο είναι το σημείο της εκκίνησης. Και θα αναφέρω κάτι πολύ συγκεκριμένο για να πλουστεύσω την κατάσταση, δηλαδή το θέμα του ότι είμαστε διαθέσιμοι για συζήτηση, βέβαια στα όρια που προβλέπονται από την εντολή που έχω λάβει, ε, μπορούμε να Έχουμε συναντήσεις, εμείς θα σας καταθέσουμε και μία αναλυτική απάντηση για τις ε, ερωτήσεις ε, και βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας ε, για να επανέλθω και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αξιολογήσουμε όχι μόνο τις ανάγκες του κοινοβουλευτισμού αλλά μπορούμε να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε μια απαρίθμηση συγκεκριμένων αιτήσεων και κατόπιν τούτου για μια ε, πιο λεπτομερή απάντηση θα πρέπει να συζητήσουμε σε μια συνεδρίαση η οποία όπως ε, καταλαβαίνετε ε, δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μία και μόνο ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τελικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο διάλογό μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε στο μέλλον σχετικά με την εσωτερική ασφάλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και λυπάμαι που καθυστερήσαμε, λιγάκι που καθυστερήσαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σε τρία-τέσσερα λεπτά. Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια παρανόηση. Σίγουρα δεν μέτραμε τα θύματα ε, της διακίνησης ανθρώπων στην Ευρώπη σε αυτούς τους 1.100. Μιλάμε για 1.100 ύποπτους εγκληματίες. Ορισμένοι από αυτούς κατηγορούνται για σημαντικές ε, ποινικέ πράξεις ε, φυσικά ακόμα είναι ύποπτοι, δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί οι υποθέσεις τους. Ε. Δέκα χιλιάδες λοιπόν ύποπτοι παράνομοι μετανάστες ελέγχθηκαν από τη Frontex σε διάφορα σημεία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών μαζί με άλλες πληροφορίες που συλλέξαμε σε αυτές τις εννέα ημέρες μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε 170 διακινητές αυτών των παράνομων μεταναστών. Οι διακινητές λοιπόν, τα δίκτυα ήταν ε, αυτό το οποίο εστιαστήκαμε στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης μαζί με άλλους 90 που διακινούσαν θύματα για σεξουαλική εκμετάλλευση στην Ευρώπη και για εργασία. Επίσης πολλοί ε, συλλήφθηκαν ε, για εγκλήματα όσον αφορά την κοκαίνη, για υποψίες ε, οργανωμένου εγκλήματος και για αυτό καταδεικνύει γιατί πραγματοποιήσαμε αυτή την επιχείρηση. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι λίστεψαν ε, κοσμηματοπολία, κατοικίες ε, σε πολλά διαφορετικά σημεία στην Ευρώπη. Είναι η τακτική τους δραστηριότητα. Με αυτή την ε, επιχείρηση που κάναμε καταφέραμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργούν αυτά τα δίκτυα συλλέγοντας πληροφορίες για το πώς συνδέονται κάποιες διαρρήξεις ε, στις Βρυξέλλες, στις ε, στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Ο κύριος Κερχόπ ρώτησε γιατί το κάναμε αυτό. Έχουμε αντιληφθεί ότι ο κόσμος του εγκλήματος έχει εξελιχθεί. Είναι πιο ενοποιημένος. Είναι πιο δύσκολο να τους αντιμετωπίσουμε τμηματικά. Δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μόνο με τα ναρκωτικά ή μόνο με την παράνομη μετανάστευση. Υπάρχουν υποδομές, δίκτυα που συνδέουν πολλές από αυτές τις εγκληματικές δραστηριότητες και ο σκοπός αυτής της επιχείρησης ήταν να προσπαθήσουμε να πλήξουμε τα κρίσιμα σημεία, τα κομβικά σημεία αυτών των δομών, αυτών των δικτύων. Στη διάρκεια της επιχείρησης καταφέραμε να συλλέξουμε πληροφορίες από έναν τομέα ας πούμε τις επιχειρήσεις που δείξαν σε συλλήψεις σε ένα άλλο τομέα με τρόπους που φαίνονται να σύνδετοι αρχικά. Καμιά φορά ασχολούμασταν με δίκτυα που, που διαπράττουν απάτες και εκεί βρήκαμε διακινητές ε, παράμων μεταναστών. Αυτό καταδεικνύει ότι πρέπει να είμαστε πιο οριζόντιοι στο έργο μας ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στη σύγχρονη φύση αυτών των ποινικών αδικημάτων. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα έχουμε με τη Frontex. Η Frontex διεξάγει αυτές τις επιχειρήσεις ε, στις κανονικές της δραστηριότητες. Μέχρι να έχουμε μία συμφωνία για τη μεταφορά δεδομένων, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ Frontex και Europol, δεν θα μπορούμε κάθε μέρα να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές με αυτόν τον τρόπο. Ανταλλάσσονται συνήθως με τις εθνικές αρχές. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Frontex και Europol στο μέλλον. Φυσικά εμείς θα εκπονήσουμε μια έκθεση όπου θα αποτυπώνονται όλα αυτά και η ερώτηση του κ. Κουάλα σίγουρα θα παράσχουμε μια έκθεση στο Κοινοβούλιο ώστε να σας πείσουμε περισσότερο για την αξία τέτοιων επιχειρήσεων. Τώρα για την ερώτηση της κυρίας ε, Λόπες για το ξέπλυμα χρημάτος, συμφωνώ. Είναι το λάδι στα εγκληματικά γρανάζια. Έχουμε ένα πλαίσιο για τις δραστηριότητες ξεπλήματος χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε είναι η πλήρης υλοποίηση αυτών των συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο. οι περιπτώσεις ε, νομοποίησης χρηματών από παρανόμες δραστηριότητες ακόμα έχουν μέλλον. Ε, χρειαζόμαστε ακόμα αρκετό δρόμο για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρο. Για να προσαρμοστεί στο χρονικό συντόμευσε αυτό που έχει να πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να δούμε τώρα αν οι συνάδελφοι έχουν κάτι άλλο το οποίο θέλουν να πούν. Ε, Μπίργκιτ, θες το λόγο. Ε, Αλλιώ θα πρέπει εγώ να κόψω από τα το πω στο μέλλον. Ε, πρόεδρε, θα ήθελα σύντομα να κάνω μια ερώτηση γιατί μιλούμε για 1100 υπόπτους. Ε, ακούσαμε. Αυτοί Εάν ήταν να τους χειριστούν οι εθνικές αστυνομίες, άραγε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα. Άρα να θεωρήσουμε ότι η Europol πρόκειται να ενημερωθεί σε σχέση με το πού κατέληξε η περίπτωση του καθενός από αυτούς, αν καταδικάστηκαν και για ποιο έγκλημα. Τώρα κάτι άλλο, όχι για τους μετανάστες αλλά για τους διακινητές αυτούς που τους βοηθούν να διασχίσουν τα σύνορα παρανόμως. Μας μιλήσατε και για διακίνηση ε, ανθρώπων. Χθες το ανέφερα αυτό εδώ στη συνεδρίασή μας. Και εσείς τι λέτε, ότι αν κάποιος ε, βοηθά κάποιον ε, μετανάστη να πάει σε κάποια ασφαλή χώρα, αυτό σημαίνει ότι είναι διακινητής προσώπων. Πρόεδρος. Δεν ξέρω κάποιος άλλος έχει κάτι να ρωτήσει συμπληρωματικά. Μόνικα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι αυτή η επιχείρηση είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό γιατί εστιάζεται στο θέμα της συνεργασίας μεταξύ των μελών και ακριβώς γι' αυτό έχουμε και την Europol. Οπότε σε αυτή τη φάση θα να σας πω ότι δεν λέω ότι η δική μου περιοχή είχε εμπλακεί στην επιχείρηση. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος στην περιφέρειά μου είχε φοβηθεί, είχε τρομοκρατηθεί από διάφορες ιστορίες που κυκλοφορούσαν. Άρα δηλαδή το θέμα των συλλήψεων δεν είναι ότι συνελήψαν εκείνοι οι οποίοι έπρεπε. Είναι πολλές φορές σε λανθασμένες περιπτώσεις. Αυτό ήταν το ένα που θέλω να πω. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επιτρέψτε μου βέβαια να το διατυπώσω, γιατί υπάρχει ένας πολύ σημαντικός στόχος πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις. Και όταν λέει κανείς κάτι, δεν θα πρέπει βέβαια να επικρίνεται για το ότι δεν υπάρχει ε, οργανωμένο έγκλημα. Το δεύτερο, εν πάση περιπτώσει, που θέλω να πω και που με ενδιαφέρει, είναι το εξής. Να δούμε ε, εφόσον ο αριθμός των αστυνομικών που είχε συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση ήταν τέτοιος που αναφέρατε εσείς πώς το κρίνετε αυτό πώς μπορεί κανείς να διαμορφώσει αυτές τις επιχειρήσεις πιο αποτελεσματικά κυρίως όσον αφορά την απόκτηση πληροφοριών από τα κράτη-μέλη δηλαδή η Ευρωπόλ παίρνει σωστή πληροφόρηση από τα κράτη-μέλη με άλλα λόγια η Europol ενημερώνεται σωστά και με τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή ήταν μία πρώτη ερώτηση. Και μία δεύτερη αφορά την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Έχω κάνει την εξής ε, εμπειρία. Ξεκινάμε από μια συμμορία αν θέλετε, αλλά υπάρχουν και διάφορες οργανώσεις όσον αφορά την παράνομη διακίνηση. Δυστυχώς σε εμά υπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρονται ως λαθρομετανάστες και μετά μεταφέρονται σε κάποια άλλη χώρα. Αυτή είναι λίγοι. Υπάρχουν όμως άλλοι, πολλοί, οι οποίοι καταλήγουν την παράνομη διακίνηση, πορνεία, ε, εμπόριο παιδιών, εμπόριο οργάνων, ανθρώπινων οργάνων, τραγικές καταστάσεις. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο ενδεχομένω υπάρχει ε, ένα συγκεκριμένο σύστημα που αντιμετωπίζει την κατάσταση και πώς συμπεριφέρονται οι οργανώσεις αυτές. Γιατί νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δομές που χρειάζεται μια κοινωνία. Κοιτάξτε. Συναδελφοί, η πρόθεσή μου ήταν ε, να απαντήσουμε αυτό που ακούσαμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ έχει ανοίξει ένας νέος γύρος ερωτημάτων. Ε, αυτό θεωρείται κακή προεδρία. Δικό μου σφάλμα. Τώρα που ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας έχει ανοίξει, οπότε αν μπορείτε να με βοηθήσετε να είστε σύντομοι και εσείς Κορνέλια Άννα Πρόσφατα ένας Κινέζος πολίτης συλλήφθηκε στην Πορτογαλία με ένταλμα σύλληψη της Ιντερπολ διότι ε, το καταζητούσαν στην Κίνα για απάτη. Είχε λάβει μάλιστα βίζα. Φανταστείτε και η πορτογαλική κυβέρνηση αρνήθηκε να μου δώσει τα ονόματα ανθρώπων που έλαβαν αυτέ τι χρυσέ βίζα για λόγου προστασία δεδομένων. Δεν ζητήσαμε καν του τραπεζικού λογαριασμού, απλά τα ονόματα. Προφανώς λοιπόν αυτό το σύστημα Golden Visa που δίνουν πολλές χώρες ε, που έχει υιοθετήσει η δική μου χώρα και που σκέφτεται να υιοθετήσει η Ιταλία είναι ένα σύστημα εισαγωγής εγκληματιών. Ό,τι καλύτερο για το οργανωμένο έγκλημα. Έχετε στοιχεία. Κάνετε κάτι για να αποθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν με αυτό το σύστημα το οποίο ουσιαστικά δεν είναι παρά ένας τρόπος εισαγωγής εγκληματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Okay, um, ο παρακαλώ, Κορνιλία. Ούτε ένα λεπτό δεν χρειάζομαι. Μιλήσατε, κύριε Ράινράιτ, κάτι για κάποια συμφωνία ε, μεταξύ Europol και Frontex, ε, με βάση κάποιες πληροφορίες. Μπορείτε μήπως ε, σχετικά με την προβλεπόμενη συμφωνία να πείτε μερικά περισσότερα στοιχεία. Δηλαδή τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να σας καταθέτουν πληροφορίες ή πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Σε ευχαριστούμε, κύριος Γιούρεκ, και κατόπιν θα, θα λάβει το λόγο ο Ρόμπιν Βουέινραϊτ. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο είναι δυνατόν να απαντήσω τώρα. Ίσως να πρέπει να περιμένω το επόμενο σημείο. Οι ομάδες διακίνησης ε, ανθρώπων, κατά την άποψή σας, είναι κινητές μονάδες. Σε ποιο βαθμό έχουν διεθνή δραστηριότητα. Είναι τοπικές ε, ομάδες που οργανώνουν τη ροή εντός μιας συγκεκριμένης χώρας προς μια άλλη ή είναι διεθνής. Πώς εκμεταλλεύονται την διεθνή κρίση για σκοπούς κέρδους μέσω της διακίνησης ανθρώπων ανοίξαμε με ένα ολόκληρο νέο γύρο ερωτήσεων, Ρομπ, ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά είμαι βέβαιο ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Ευχαριστώ. Wainwright. Ξεκινώ με την ερώτηση όσον αφορά του διακινητέ. Ήταν εύκολη ερώτηση. Από του 170 που συνελήφθησαν, έχουμε αρκετέ πληροφορίε για να δούμε σε ποιο βαθμό αυτοί είναι οι θύνοντες ε, αυτών των συμμοριών. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον θα μας ενημερώσουν για το τι έγινε όταν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία. Έχω να σας πω ότι η απάντηση είναι καταφατική και ακριβώς ε, θεωρούμε ότι ακόμα η Europol ε, δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα μπορούσε να είναι, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Και αυτό το λέω και επαναλαμβάνω συνεχώς. Έχουμε αυτή την τεράστια επιχείρηση. Έτσι θέλουμε το σύστημα να το αναγκάσουμε το ΣΥΠΗΝ να μας οδηγεί σε περισσότερη ροή πληροφοριών και να έχουμε ε, καλύτερη απόδοση στην δουλειά μας. Το είπε και ο κύριος Κέρκο, αν μπορούμε να είμαστε έτσι κάθε μέρα. Όχι, δεν μπορούμε. Θα βρούμε μια φυσιολογική ροή εργασίας, αν έχουμε και αποτελεσματική ροή πληροφοριών. Και ε, τελικά έχουμε μικρότερες επιχειρήσεις και έχουμε πιο σημειακή εστίαση της προσοχής μας όπως ας πούμε το κυβέρνο έγκλημα όπως αναφέρθηκε και θα συζητηθεί και σήμερα το πρωί κι άλλο είναι η κυρία Γκόμες για αυτές τις ε, χρυσές θεωρήσεις διαβατηρίων θα πρέπει να συζητηθεί αυτό με τις ε, αρχές της χώρας σας είναι καινούριο, δεν το ήξερα το θέμα θα το λάβω υπόψη. Ένστ, ε, αναφέρατε για τη συμφωνία μεταξύ Frontex και Europol προβλέπεται στον κανονισμό για την Frontex το ότι θα μπορεί να, να στέλνει στην Europol σε συγκεκριμένα πλαίσια μη επεξεργασμένα δεδομένα ούτω ώστε και εμείς να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για να βοηθάτε το έργο μας και έτσι να μπορούμε να χτυπήσουμε τους ε, διακινητές. Όσον αφορά τα ποσοστά που είπατε κύριε Γιούρεκ, έτσι γίνεται με το οργανωμένο έγκλημα. Είναι όλο ένα και πιο διεθνής, είναι πιο ευκίνητη ας το πούμε, πιο ευέλικτη αυτή οι εγκληματίε. Συνεργάζονται βέβαια και με τους τοπικούς διακινητές, αλλά έχουμε και κάποιες συμμορίες που έδρασαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλες τις χώρες. Τώρα τι γίνεται με, με την κατάχρηση των ελευθεριών που έχουμε για το ίντερνετ, τη διακίνηση, για την ε, παγκοσμιωμένη κοινωνία, ε, το κάνουν αυτό, ναι, ούτως ώστε να έχουν ένα πλεονέκτημα. Άρα και εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε με κάποιο, πάλι σε επίπεδο διεθνές, σε επίπεδο ολοκληρωμένο, σφαιρικό. Ρόμπλε, πρώτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε που έμεινες μαζί μας για να απαντήσεις σε αυτές τις επιπλέον ερωτήσεις. Με μεγάλη μας χαρά, ας ξαναδούμε. Σε λίγο θα μας μιλήσεις για το κυβερνό που είναι το επόμενο θέμα της μέσα διάταξης. Και τώρα, κοιτάξτε, το επόμενο επόμενο, είναι θέμα ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων. Υπάρχει αυτή η προφορική ερώτηση με συζήτηση. Προβλέπεται για την Ολομέλεια και αφορά την εσωτερική ασφάλεια. στη ΛΥΜΠΕ. Θα ψηφίζουμε σε σχέση με την στατική ιστορική ασφάλεια και οι συντονιστέ το συζητήσουν ακριβώ όπω κάναμε για την Μεσόγειο. ίδια μέθοδος εργασίας όπως και για την Μεσόγειο και να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα οποία προτείνουμε για στρατηγική ιστορία ασφάλειας για τα βασικά θέματα αυτής πρόκειται να τα προωθήσουμε όπως πρέπει. Αν θέλει κάποιο να πει κάτι, προχωρούμε. Αυτό το είπα απλώς ενημερωτικά. Συνάδελφοι. Μία ερώτηση για αυτό, για την με την προφορική ερώτηση. Ναι, εντάξει. Ε, έχετε το λόγο. Weinberg. Έχετε, ε, μας τελειώσετε την ενημέρωση. Ναι, ναι, ναι, ρωτήστε, τέλειωσα την ενημέρωση. Ωραία, λοιπόν, θα την κάνω στα σουηδικά. Έχω μια ερώτηση για το τι συμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κίνδυνος εδώ να τολμήσει να εφαρμόσει μια στρατηγική η οποία μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική. Γιατί εμεί είχαμε τρεις ε, Σουηδούς που έρχονταν από τη Σομαλία σε εμά, οι οποίοι ε, αξιοποίησαν, εκμεταλλεύτηκαν διάφορους κανόνες που υπάρχουν και ό,τι γίνεται εκεί στη Σομαλία και ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Έχουμε βέβαια πολλές συμφωνίες, το ζήτημα του ανοίγματο των συνόρων. Ένας από αυτούς είχε τη δυνατότητα να πάει στη Συρία όπου συμμετείχε σε δραστηριότητες ε, δουλείας, ε, βίας. Αυτά τα τρία μέλη της ΑΣΥΣ κατάληξαν να έχουν σοβαρά προβλήματα και τα πράγματα επιδεινώνονται κιόλας διότι υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει περίπτωση να κάνουν εγκληματικές πράξεις σε κάποιο εμπορικό κέντρο στη Σουηδία. Τίθεται λοιπόν το ζήτημα της ασφάλειας και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσαμε να αποφύγουμε τέτοιου είδου καταστάσεις ε, προβλήματα στη Σουηδία και αλλού στον κόσμο. Τι θα κάνετε για να αποφύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα αντιπαραγωγικά που σε πολιτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Ε, οι συναδελφοί μου προετοιμάζουν την προφορική ερώτηση, οπότε θα χρειαστεί να στείλετε τις ερωτήσεις σας μέσω του συντονιστή σας. Αυτό είναι το σημαντικό. Και η συζήτηση θα γίνει στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια Στείλτε λοιπόν την ερώτηση έτσι για να μην ξεκινήσουμε εδώ τη συζήτηση στην Επιτροπή διότι ε, θα πρέπει να το συζητήσετε με του συντονιστέ σα. Ευχαριστώ. Okay, colleagues, if there are no other points of... Αν δεν υπάρχουν άλλα ενημερωτικά σημεία ή ερωτήσει, θα περάσουμε αμέσω στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την παρουσίαση τη αξιολόγηση του κινδύνου που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα που διευκολυνείται από το διαδίκτυο και να ευχαριστήσω τις για τις σχετικές ερωτήσεις. Η παρουσίαση από τον κύριο Wright, διευθυντή της Ευρωπόλ, Ρομπ. Στρέφομαι απευθείας σε εσά για την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ. Και πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για αυτό το σημείο είμαι ο μόνος ομιλητής, οπότε να έχω περισσότερο χρόνο και βέβαια θα κάνουμε ό,τι πει ο Πρόεδρος και για να έχουμε χρόνο ε, να περισσέψει χρόνο τέλο πάντων για τις ορκές από τους βουλευτές. Ο βασικός στόχος αυτής της συνάντηση είναι να ανταλλάξουμε απόψεις όσον αφορά το κυβερνό έγκλημα ε, και, και κυρίως στα πλαίσια αυτής της έκθεσης που δημοσιοποιήσαμε. Έχετε εδώ αυτό το φυλάδιο, ο κύριος Άλμπεχτ αναφέρθηκε σε αυτό Οπότε πρόκειται επομένω για την αξιολόγηση του 2014 για το κυβερνοέγκλημα ε, από το κέντρο κυβερνοεγκλήματος της Europol που ξεκίνησε το 2013 τις εργασίες του. Και αυτό αφορά τους νομοθέτες, τους ασκούντες στην πολιτική, ε, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις σχετικές απειλές. Έχουν βοηθήσει οι διευθυντικές αρχές από όλες τις χώρες μέλη, αλλά και από πανεπιστήμια και από τον ιδιωτικό τομέα. Να σας πω ε, τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης, αλλά επίσης να σας πω από την εμπειρία μου τι γίνεται για ορισμένα ζητήματα ε, τα οποία θα είναι ενδιαφέροντος και αρμοδιότητό σας. Πρώτα-πρώτα δύο λόγια για το κέντρο κυβέρνου εγκλήματος στην ε, Europol. Βολεύουμε το σύνδεσμο ε, μοντέλο για τις δυνατότητές μας όσον αφορά τις πληροφορίες για το συντονισμό και γι' αυτό και έχουμε τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών, έχουμε πάνω από 100 αναλυτές και κάθε μέρα αναλύονται οι πληροφορίες και έχουμε 160-170 αξιωματούχους συνδέσμους για να συντονιζόμαστε με τις εθνικές διοικητικές αρχές. Οπότε και σε αυτό το σημείο έχουμε μια πλατφόρμα συντονισμού, έχουμε ένα κόμβο συντονισμού για το θέμα της αντιμετωπίσης του γεγονέγκληματος, ασφαλές περιβάλλον με αναβαθμισμένη προστασία και έχουμε τις συνήθεις, ε, συνήθεις διαδικασίες Όλα αυτά γίνονται το 2013 και έχουμε επομένως ε, τρία μέτωπα. Πρώτα πρώτα ε, απάτες από το ίντερνετ. Έχουμε επίσης ε, για ναρκωτικά, λαθρέα και όπλα. Το λαθρεμπόριο που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο από αυτούς τους κυβερνοεγκληματίες. Να πάρετε επομένως μια ιδέα. Είχα μια στατιστική της ECB ότι η απάτη φτάνει σε κύκλο εργασιών πάνω από 1,3 δις ετησίως. Είναι η απάτη από το ηλεκτρονικό εμπόριο που συνεχώς ε, φουσκώνει όσον αφορά τις συναλλαγές που κάνουν οι καταναλωτές μέσω του ίντερνετ. Τώρα όσον αφορά την μετάλλευση ανηλίκων και εδώ ασχολούμεθα πολύ γιατί η κλίμακα του προβλήματος είναι μεγάλη, μεγάλη η διαστροφή τελικά που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και έχουμε πέντε μέτωπα για τα δίκτυα, ε, έχουμε χιλιάδες ε, προσώπων που συμμετέχουν στο, στο υλικό που προκύπτει από την ε, κακοποίηση των υλίκων, εκατοντάδες είναι οι ύποπτοι, από τις λίγες υποθέσεις λείψαμε φέτος 15 ειδικοί από 8 χώρες συνεδριάζουν στην Europol και έχουμε μέσα αυτή την task force για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε 4 εκατομμύρια ε, περιπτώσεων ε, κακοποίησης ε, ανηλίκων. Ε, μιλούμε για φωτογραφίες, για φιλμ. 5 ε, τεραμπάιτ είναι το όγκος αυτών των δεδομένων. Και βεβαίως όλοι αυτοί οι μας βλέπουν φρικτές εικόνες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο είναι αυτό το φρέσκο υλικό το οποίο συνεχώς ανεβαίνει στο διαδίκτυο και βλέπουμε μέσα ένα και περισσότερη βία που έχει να κάνει με την σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων. Αλλά βέβαια επίσης όλο ένα και πιο μικρά παιδιά αφορά αυτή η κακοποίηση. Το 10% είναι κάτω από 2 ετών. Διαπιστώσαμε επίσης στο μεταξύ Έχουμε λένε και περισσότερη κρυπτογράφηση από πλευρά αυτών των δικτύων για να κρυφτούν τι οι ε, δραστηριότητε αυτές. Έχουμε επομένω και εμείς ε, του καλύτερους ε, ειδικού για πληροφορική. Έχουμε σκληρούς δίσκους που τους έχουν τώρα οι, οι ερευνητές και προσπαθούν να ανοίξουν κάποιους από αυτούς που είναι δύσκολο γιατί ακριβώς την κρυπτογραφημένα τα δεδομένα. Ε, επίσης έχουμε και κάποιες κυβερνοεπιθέσεις για την ε, υποδομή και άλλα θέματα ε, όπως όπως, την υποκλοπή κωδικών τραπεζικών λογαριασμών και τέτοιες δραστηριότητε. Προσπαθούμε επίσης να ελέγξουμε την κατάσταση και τους ιούς αυτούς που φτιάχνουν στα πλαίσια της εγκληματικής δραστηριότητα. Τώρα προσπαθούμε να δούμε αυτοί οι hackers πόσο βλάπτουν τις οικονομίες. 300 δις δολάρια ετησίω λένε ότι είναι το πλήγμα της οικονομίας. 50 έρευνες έγιναν τελευταίο χρόνο. επίσης προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά της κρυπτογράφησης στα εργαστήρια από τους ειδικού μας, από τον δυτικό τομέα, την πληροφορική, πανεπιστημιακούς κλπ. Όλο και περισσότερο με τον ιδιωτικό τομέα και το πανεπιστήμια έχουμε δύο ε, ομάδες ε, εξειδικευμένες και έχουμε υπογράψει μνημόνιους συνεννόησης με δέκα εταίρους εστιαζόμενοι στο μέγιστο δυνατό βαθμό στο να έχουμε επιχειρησιακά αποτελέσματα. Τους πρόσωπους μήνες συστήσαμε μια task force για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο με τους πιο τακτικούς συμμετέχοντες των κρατών μελών. Η δουλειά μας επίσης μας επιτρέπει να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα των στρατηγικών τάσεων του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο το οποίο μας επιτρέπει να εκπονήσουμε αυτή την αξιολόγηση απειλών που βλέπετε. Κάλυψα ήδη κάποια πτυχές στην εισαγωγή μου. Δύο-τρία οριζόντια ζητήματα που συνδέουν μεταξύ τους τα εγκληματικά προβλήματα online είναι ότι το δήμα στον κυβερνό χώρο αυξάνεται, γίνεται πιο εξειδικευμένο και σίγουρα αυξάνεται και ο αριθμό επιθέσεων και η τάση που παρατηρούμε είναι μια, η ανάπτυξη μιας ε, εγκληματικής βιομηχανίας βασισμένης στις υπηρεσίες. Όλο και περισσότερες ε, εγκληματικές ομάδες μπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες απασχολώντας εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, εργαλείων και ε, υπηρεσιών. Για λίγες εκατοντάδες ευρώ κάποιος μπορεί να νοικιάσει ένα botnet για να ξεκινήσει μια εκστρατεία spamming κατά ενός ανταγωνιστή ή για να διανύμει ένα malware. Ένα botnet μπορεί να σπάσει κωδικούς, να βοηθήσει να κλέψουμε στοιχεία τραπεζικών δεδομένων, ε, να κλέψουμε ταυτότητα. Είναι πολύ εύκολη η διάπραξη ε, εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και η ποικιλομορφία των δραστών ε, δείχνει πως μεγάλη ανάγκη υπάρχει να το αντιμετωπίσουμε. Τα κέρδη φυσικά είναι τεράστια και αυτό οδηγεί σε αυτή την τεράστια επέκταση του προβλήματος του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Οι παραδοσιακές ε, εγκληματικές ομάδες ε, διευρύνονται, προσλαμβάνουν πτυχιούχους για να πουλήσουν ναρκωτικά, για παράδειγμα, ή επενδύουν σε νέες μεθόδους. Πρόσφατα νοικιάζουν ή αγοράζουν botnet χρησιμοποιώντας malware που κλέβει ένα ευρώ από ένα εκατομμύριο τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη. Είναι σχεδόν αδύνατο να ανοιχνευτεί τόσο από τα θύματα ή από, ούτε, όσο και από τις τράπεζες. Η απο οσο και απο τις τραπεζες η εκθεση μας δείχνει επίσης μεταβολή στον τρόπο αλληλεπίδραση μεταξύ των εγκληματιών. Παραδοσιακά οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος χαρακτηρίζονταν από βιοπραγίες μεταξύ τους. Ε, ε, αυτός ο βίος ανταγωνισμός έχει αντικατασταθεί από ένα πιο συνεργατικό περιβάλλον. Τώρα στον κυβερνοχώρο οι εγκληματικές ομάδες ε, λειτουργούν περισσότερο ως επιχειρησιακοί εταίροι παρά ως ανταγωνιστές. και παρατηρείται μεγαλύτερη οργάνωση και διάρθρωση που μπορεί να εξελιχθεί και στο μέλλον. Σημαντικά ζητήματα τίθενται όσον αφορά την εξέλιξη της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και του ρόλου της αστυνομίας ε, στις online τεχνολογίες. Όλα έχουν φυσικά αλλάξει πολύ. Όλοι περνάμε ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας online ε, σε καταστήματα, στο υπολογιστικό νέφος και τα λοιπά. Δεν θα σας εκπλήξει ότι και οι εγκληματίες πλέον χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τα εγχειρήματά τους. Λειτουργούν από χώρε που συχνά δεν συνεργάζονται μεταξύ τους, καταχρώνται των ε, τεχνολογιών κρυπτογραφής για να παραμένουν κρυφοί, αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται όλα τα κενά στις εθνικές νομοθεσίες για να αποφύγουν τη δίωξη, κερδίζοντας εκατομμύρια ευρώ εις βάρος των επιχειρήσεων και των πολιτών μας. Πολύ απλά οι δυνατότητες των αστυνομικών δυνάμεων δεν είναι επαρκής ε, για να αντιμετωπίσουν τις ταχαίως εξελισσόμενες αυτές απειλές. Ένας λόγος είναι ότι οι αστυνομίες πρέπει να αναπτύξουν τις ψηφιακές έρευνες ε, και να αποτελέσουν αυτές ε, βασικό κομμάτι της εργασίας τους. Πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της αστυνομικής συνεργασίας και των σχετικών μηχανισμών. Κάτι που αναφέραμε στην προηγούμενη παρουσίαση στο πλαίσιο της επιχείρησης Αρχιμίδης και πρέπει να εμπλέξουμε και τη βιομηχανία περισσότερο και στους τρεις τομείς αυτούς που είναι δύσκολοι η Ευρωπόλ προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τα πράγματα αλλά υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο δεν έχει Ευρωπόλ άμεσο έλεγχο και είναι εξίσου σημαντικό είναι ο βαθμός στον οποίο η νομοθεσία δεν συμβαδίζει με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και αυτό υποβαθμίζει τις δυνατότητες ε, της αστυνομίας. Ε, δεν μπορούν ε, οι δυνατότητες της αστυνομίας στον πραγματικό κόσμο να αναπαραχθούν στον ψηφιακό κόσμο και πιστέψτε με υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο όσον αφορά τις ικανότητες των αστυνομικών δυνάμεων να μας διατηρήσουν ασφαλείς. Όσον αφορά την ανομιμία που έχουμε όλοι online, απολύτως νόμιμο, κανείς δεν θέλει να το αλλάξει αυτό, Παρατηρούμε όμως ότι και εμπορική παροχή υπηρεσιών όπως η Google χρησιμοποιούν ε, δεδομένα προσωπικά για να δείξουν διαφημίσεις. Η Amazon προβλέπει τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές μελετώντας τη βιβλία έχω αγοράσει τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι ειρωνικός αυτός ο δημόσιος διάλογος ε, μετά την υπόθεση Snowden όταν έχουμε τέτοιους παρόχους υπηρεσιών τόσο αεροπορικές εταιρείε που διατηρούν στοιχεία και δεν επιθυμούμε να τα διατηρούν οι αστυνομικέ αρχέ, αλλά φυσικά όπω και εσεί ε, εκτιμώ το απόρριτο, την ιδιωτικότητα, εκτιμώ το έργο πολλών και εδώ στο Κοινοβούλιο για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του πακέτου προστασία δεδομένων. Είναι κομμάτι των θεμελιωδών ελευθεριών και το δέχομαι και Πράγματι στην επιβολή του νόμου ίσως πρέπει να πάμε λίγο πιο πέρα από τους εμπορικούς παρόχους υπηρεσιών για να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λειτουργούμε με διαφάνεια ώστε να μας εμπιστεύεται το κοινό. Σημαίνει ότι πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα στον Ευρωπαίο πολίτη τι απειλές έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όχι γενικά, αλλά πολύ συγκεκριμένα, με λεπτομέρειες. Σήμερα οι εγκληματίες χρησιμοποιούν νόμιμες ε, τεχνικές κρυπτογράφησης για να κρύβονται online. Όπως γνωρίζουμε στον τομέα του Darknet, ε, το κομμάτι που δεν ε, εμφανίζεται με τους μηχανισμούς αναζήτησης. Έτσι επικοινωνούν μεταξύ τους με διάφορες τεχνικές και φυσικά όλοι όσοι βρίσκονται στο Darknet δεν είναι εγκληματίες αλλά κάποιοι έχουν συσταθεί με εγκληματική πρόθεση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, ένα παράδειγμα είναι η ανταλλαγή υλικού σεξουαλικής ε, εκμετάλλευσης παιδιών. Το 2014, για να σας δώσω μια εικόνα, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια χρήστες του το εκ των οποίων ένα τρίτο διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούν το ΤΟΡ και σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο φέτος, σε διάστημα μιας εβδομάδα, το 20% αυτών των ιστοσελιδών σχετίζονται με σεξουαλική ε, εκμετάλλευση παιδιών. Ένα άλλο 20% πουλά ναρκωτικά και ένα 40% σχετίζεται με κλεμμένα στοιχεία πιστοτικών καρτών. Πάνω από το 50% λοιπόν των φόρουμ και των ιστοσελίδων στο ε, σκοτεινό δίκτυο, στο Dark Network, ε, αφορά παράνομες δραστηριότητες και αυτό είναι σημαντικό κομμάτι που χαρακτηρίζει τη φύση του Tor Network. Ε, ταυτόχρονα φυσικά Υπάρχει και ένα σημαντικό ζήτημα. Δεν θέλουμε να καταπιέσουμε την ελευθερία λόγου. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι το TOR για τους ε, αντιφρονούντες, για τους πολιτικούς αντιφρονούντες σε διάφορες χώρες στον κόσμο. Και σίγουρα εγώ δεν πρόκειται να ζητήσω προσωπικά τέτοια αλλαγή, αλλά πιστεύω ο ρόλος μου ως εκπρόσωπος των αρχών τη τάξης, πρέπει να σας πω ότι στο μεταξύ το δίκτυο TOR διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό σοβαρά εγκλήματα και την εξέλιξη της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. Η ανωνυμία δεν μπορεί να σημαίνει ατιμορρησία. Πρέπει οι αρχές ε, της τάξης να μπορούν να προσδιορίσουν ποιος βρίσκεται online και να μπορούν να αναχαιτήσουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, φυσικά όταν αυτό αιτιολογείται λόγω ευλογών υποψιών και υπό την απαραίτητη δικαστική επίβλεψη. Η αρχή λοιπόν της νόμιμης αναχέτησης των επικοινωνιών πάντα ήταν δεκτή στην Ευρώπη και χρησιμοποιείται από τις αρχές επιβολής του νόμου με κανονικό τρόπο με επαρκή μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας των πολιτών. Μιλάμε εδώ για την παρακολουθή τηλεφωνικών επικοινωνιών που είναι κλασική τεχνική αστυνομική υπό την κατάλληλη δικαστική επίβλεψη. Δεν θα πρέπει να είναι διαφορετικά τα πράγματα online, αλλά είναι και οι ιδιωτικέ αρχέ προσπαθούν έτσι να δουν τι γίνεται όσον αφορά κάποιε κάποιες στο δίκτυο που διευκολύνουν τελικά του εγκληματίες γιατί έτσι βλέπουμε πως το ίντερνετ γίνεται ε, ε, ένας ασφαλής χώρος και τελικά όλοι εκεί πέρα αναπτύσσουν μια καθημερινή φυσιολογική δραστηριότητα. Έχουμε βέβαια την αρχή της ελευθερίας του λόγου να τη σεβαστούμε αλλά επίση θα πρέπει να προστατεύσουμε την ασφάλεια του κόσμου Όσο αφορά το ίντερνετ. Για να δούμε τώρα. Και όπως είπαμε, έχουμε το εργαστήριο, προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, προσπαθούμε να συντονίσουμε όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις. Είδατε και την Παρασκευή τα αποτελέσματα αυτής της τελευταίας επιχείρησης και εκεί συντονίσαμε 16 χώρες και τις είπα. Εκεί επισημάναμε ε, και κλείσαμε 410 ε, σκοτεινά ε, websites για ναρκωτικά, για τραπεζικά στοιχεία. Γίνανε 17 συλλήψεις επίσης, έχουμε κατασχέσει πολλά χρήματα και ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Είναι εγκληματικά site επομένως δεύτερης γενιάς και τον διαχειριστή τον ε, συλλάβαμε οπότε προσπαθούμε να δούμε ποιοι είναι κάθε φορά οι διαχειριστές αυτών των ε, ιστοτόπων και γίνεται αυτό και με παραδοσιακή παλιωμοδίτικη αστυνομική μέθοδο. Έχουμε επίσης και κάποιους ε, αστυνομικού οι οποίοι αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και μας παρέχουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες αντίστοιχα τη δράση του Και αυτές είναι οι προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσουμε ε, όσον αφορά το τοπίο της εγκληματικότητα και το τι γίνεται με το οργανωμένο έγκλημα. Ε, Βεβαίω, στο μεταξύ, οι συνομοθέτες και δύο τώρα το Κοινοβούλιο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να μας δώσουν τα απαραίτητα εργαλεία. Ε, πρώτα-πρώτα, για παράδειγμα, θα πρέπει να έχουμε πρώτο χέρι πληροφορίες, για το 85% των σχετικών ε, πληροφοριών την ε, πληροφορική αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και επομένως αφορά τον ιδιωτικό τομέα του τι γίνεται στο ίντερνετ και αντίστοιχα ο ιδιωτικό τομέα μας δίνει τι πληροφορίε για να χτυπήσουμε την και έχει η, ε, η Microsoft κάποια botnet δικά τη και αυτό και λειτουργεί η Microsoft παράλληλα με εμάς. Δεν είναι σωστό αυτό, αλλά ε, έτσι γίνεται. Έτσι, έτσι γίνεται η κατάσταση, έτσι διαμορφώθηκε η κατάσταση στο ίντερνετ. Βλέπετε επομένω την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με τι διοικητικέ αρχέ. Άρα θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό επίση αφορά και την οδηγία τη νίκαια που σήμερα, θα, αυτή τη βδομάδα, θα ζητηθεί σε τριμερή διάλογο και έχουμε κάποιο είδου ε, διαρροέ. Ε, άρα θα πρέπει να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους εμπειρογνώμονες, αυτοί που μελετούν τις, τις επιθέσεις. Επίσης η Κομισιόν έχει πει ότι πρέπει αυτές οι πληροφορίες να ανταλλάσσονται με τις διοικητικές αρχές, ιδίως ε, με την ε, υπηρεσία της Europol και κάθε τέτοια διαρροή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Άρα είναι σαν, όπως λέμε, θα πρέπει να έχουμε καλή κλειδαριά στην πόρτα για να μας διαρρήξουν, ε, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και η αστυνομία να συλλάβει τους διαρρήκτες αλλιώς θα ξαναγυρίσουν για διάρρηξη και με, καλύτερη μέθοδο. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει, να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά ε, τη, τις, και αυτά που προσπαθεί να ρυθμίσει η σχετική οδηγία. Έχουμε τους εμπειρογνώμονες ε, οι οποίοι εξετάζουν τα τεχνοκρατικά ε, ζητήματα και μας ενημερώνουν ε, όπως και εμείς ασχολούμαστε με τους εγκληματίες. Τον κύριο Σουβάβ τη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας καλώ να τους υποστηρίξετε αυτή τη βδομάδα που θα γίνει ο τριμερής διάλογος. Επίσης έχουμε αυτό το σχέδιο κανονισμού και θα συνεργαστώ από αυτό με τον κύριο μέρα Και υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διάταξη που τη διέγραψε το Κοινοβουλίο και θα μας εμποδίσει τη δουλειά μας, δηλαδή του να επιτρέπουμε σε ιδιώτες εταίρους ε, να έχουν και αυτή πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες όπως η Europol και η διεθνή Αστυνομία. Και θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί αυτά είναι σημαντικά. Ας πούμε το Google έχει βάση στην Ιρλανδία και μία από τις υπηρεσίες τους είναι ότι θα μπορούσαν να βρουν ε, τις πιστατικές κάρτες ε, που διατρέχουν κίνδυνο. Και θέλουν αυτό, ας πούμε, να το κοινοποιήσουν να βρουν τους κατάλληλους ε, συνδέσμους. Είναι σαφές ότι στην Ευρώπη έχουμε κοινή αγορά και ένα σημείο διέλευσης μπορεί να ε, προκαλέσει πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά με βάση αυτά που σκύνει για τη Europol, η Google δεν μπορεί να στείλει αυτά τα στοιχεία άμεσα στη Europol. Είτε θα πρέπει να τα πουλήσει στο κράτος μέλος των ιδιοκτητών και στα 28 αν θέλετε ή όλα θα πρέπει να τα περάσει από τη Europol της Ιρλανδίας ε, που είναι μία από τις μικρότερες ε, και λιγότερο εξοπλισμένες στην Ευρώπη. Άρα τι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν ούτε οι πόροι ούτε οι δυνατότητες. Και με τον τρόπο αυτό οι εγκληματίες ε, συνεχίζουν ανενόχλητη τη δράση τους. Υπάρχει εδώ μία απλή λύση, δηλαδή να επιτραπεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε πολίτες να έρχονται και αυτοί σε επαφή με τη Europol όπως ισχύει ε, και με όλους τους άλλους οργανισμούς. Βεβαίω, και έχουμε και τον τεχνικό εξοπλισμό και το πλαίσιο προστασίας δεδομένων και νομίζω ότι απλά πρέπει να βελτιωθούμε στον τομέα αυτό, στο μέλλον. Τελειώνω με ένα τρίτο παράδειγμα που και πάλι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, την οδηγία περί κατακράτησης ή μάλλον απόσυρσης δεδομένων. Και εδώ ο στόχος της διατήρησης των δεδομένων είναι ε, γιατί εξυπηρετεί την δημόσια ασφάλεια. Βέβαια έχουμε ανησυχίες σχετικά με το ότι ε, αυτή η οδηγία μπορεί να πάψει να ισχύει χωρίς τη διατήρηση, την ε, διαφύλαξη των ε, δεδομένων νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε τελικά να είμαστε επιτυχημένοι σε αυτό τον τομέα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ τα δεδομένα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον, στην αντιμετώπιση των εγκληματιών γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η σχετική οδηγία θα αντικατσαθεί από ένα αποτελεσματικό νέο μέσο που Βεβαίως ε, δεν θέλω εδώ να μπω σε χωράφια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως το ίδιο θα ήθελα να πω και για την ε, αρχή περί υποκλοπής επικοινωνιών η Google, παραδείγματος προσπαθεί να έχει μηχανήματα αποκρυπτογράφησης και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη σε ένα τομέα όπου ο ιδιωτικός τομέας εργάζεται με το δημόσιο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι προσπάθησα να σας παρουσιάσω με ειλικρίνεια τις απειλές από το κυβερνοέγκλημα και υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί ευαίσθητοι τομείς. Ε, εγώ δεν ήρθα εδώ με πολιτικό θεματολόγιο, μιλάω ως άνθρωπος της πράξης και ως άνθρωπος της ε, πράξης ε, πρέπει να σας πω ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εκπροσωπώ σωστά την, ε, τον φορέα μου και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη. Βεβαίως ο νομοθέτης, το κοινοβούλιο αν θέλετε, καλείται να αποφασίσει πόσο πιο πολύ μπορεί να προχωρήσει ο νομοθέτης για να διαφυλάξει το νομοθετικό περιβάλλον, να ε, επιφέρει και να αναπτύξει ε, νομοθετική δραστηριότητα με ισορροπημένο τρόπο. Η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αποφύγει τη συζήτηση για ένα δίλημα που προκύπτει από τις πολύ εξελιγμένες ε, τεχνικές ε, κρυπτογράφησης ε, που χρησιμοποιούνται και κωδικοποίησης. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις, δραστηρι... τις αρμοδιότητές μας και επιγραμμικά και να βρούμε ένα σύστημα το οποίο προσφέρει η Χέγγε. Υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις και αυτή τη συζήτηση πρέπει να την έχουμε με ειδικού της πληροφορικής, της προστασίας δεδομένων, της επιβολής του νόμου για να καταλήξουμε στη σωστή λύση. Με, μια θετική, ε, με ένα θετικό συμπέρασμα καταλήγω, να αξιολογήσουμε τις ε, προκλήσεις από το κυβερνό έγκλημα. Αυτό είναι θετικό γιατί μόνο τώρα που το αξιολογούμε το πρόβλημα μπορούμε να εντοπίσουμε την κλίμακά του και το τι πρέπει να γίνει. Και έτσι λοιπόν ε, Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας, για τη σύσταση και τη χρηματοδότηση του Κέντρου Κυβερνοεγκλήματος. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς την υποστήριξή σας. Και επιπλέον θέλω να σας ευχαριστώ και για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε κυρίως με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για όλα αυτά τα περίπλοκα θέματα. Και όπως πάντα θέλω να κλείσω υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος της ε, Europol είναι να λειτουργεί με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Πολλοί από εσά έχετε έρθει στην Χάγη, αλλά απευθύνω την πρόσκλησή μου κυρίως στα νέα μέλη για να δείτε τι ακριβώς κάνουμε. Ελάτε να μιλήσετε με τους υπευθύνου ε, προστασίας δεδομένων ε, και με τους εκπροσώπους εθνικών αστυνομιών που έχουμε εμείς στην υπηρεσία μας. Μα Κρηγόρησα κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ όμως που με αφήσατε να τελειώσω την, και να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίτηδες αφήσαμε πολύ χρόνο για αυτό το θέμα σήμερα, γιατί νομίζω ότι στο τέλος ε, της ομιλίας σας είπατε ότι τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα, αλληλένδετα και πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι τα θέματα του ε, κυβερνοεγκλήματος ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλους ενδιαφέρουν τους ε, συναδέλφους και έχουμε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για όλα αυτά γιατί σας είπα είναι ελένδετα τα θέματα και μας ε, απασχολούν ε, σε σχέση με, την, με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο, με την κωδικοποίηση θέματα που συνδέονται μεταξύ τους. Αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές ε, προκλήσεις. Ε, καλούμε να αντιμετωπίσουμε το κυβερνοέγκλημα και να προστατεύσουμε όμως και την ιδιωτική σφαίρα. Ε, μεγάλες οι προκλήσεις για μας, για την Επιτροπή μας. Έχουμε χρόνο για συζήτηση, αρκετό χρόνο. Σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Wainwright για την παρουσίαση αυτή και για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι πολύ σημαντικές. Ε, χρειάζεται να εντείνουμε την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ειδικότερα και το οργανωμένο έγκλημα στο διαδίκτυο. Συμφωνώ απόλυτα και θαυμάζω το έργο της Ευρωπόλ και ειδικά του κέντρου εγκλήματος στον κυβερνοχώρο για την Ευρώπη και πιστεύω ότι πρέπει να έχει κοινέ ερευνητικέ ομάδες και χρηματοδότηση. Το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά διότι αυτοί διενεργούν τις έρευνες των υποθέσεων και εκεί έχετε την πλήρη μας υποστήριξη. Όσον αφορά την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, να σας πω μια ιστορία. Κοιτώντας ε, τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία για τα εγκλήματα, το ποσοστό περιπτώσεων βίας κατά γυναικών και ανηλίκων κυρίως λαμβάνει χώρα σε οικιακό περιβάλλον, εντός οικογενειών, εντός κατοικιών και νοικοκυριών. Εγώ λοιπόν στη θέση σας θα ακολουθήσω την ίδια διαδικασία που προτείνεται για την κρυπτογράφηση. Θα έλεγα ότι οι αρχές ε, ε, επιβολής του νόμου, οι αστυνομικέ αρχές, πρέπει να ρίξουν μια ματιά στα πίσω δωμάτια των ε, οικογενειών. Φυσικά θα διαγράψουμε όλα τα βίντεο, όλα τα δεδομένα, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα αλλά για λόγους πρόληψης της βίας ε, σε αυτούς τους χώρους. Γιατί εκεί συμβαίνει στο μεγαλύτερο ποσοστό. Ναι, μπορεί κανείς βέβαια να ισχυριστεί το αντίθετο. Μπορεί να ισχυριστεί ότι σήμερα μια αστυνομική αρχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όταν συναντώνται εγκληματίες ε, του οργανωμένου εγκλήματος κάπου στο δάσος, κάπου όπου δεν περνάνε συνήθως αστυνομικοί. Οπότε εκεί δεν μπορεί κανείς να ξέρει πού θα συναντηθούν κάτω από κάποια γέφυρα, κάπου αλλού. Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα πρέπει να καταχωρούμε το πού πηγαίνει ο καθένας μας, ώστε να γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο καθένας και έτσι να μπορούμε να εντοπίσουμε εγκληματίες, να μπορούμε να τους παρακολουθούμε. Για όλους. Ε, όσοι δεν χρειάζεται να κρύψουν τίποτα, τα δεδομένα τους μπορούν να διαγραφούν. Η ερώτηση είναι λοιπόν γιατί δεν το κάνουμε. Question is, why don't we do that? Γιατί δεν το κάνουμε. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθούσε εντυπωσιακά να εντοπίζουμε το οργανωμένο έγκλημα στην πραγματική ζωή, όπου οι ευκαιρίες να παρακολουθούμε τις κινήσεις του καθενός είναι τόσο λίγες. Ενώ στο διαδικτυακό περιβάλλον όλοι παρακολουθούνται με τη βοήθεια της υποδομής, των διευθύνσεων IP κτλ. Να σας πω γιατί. Λόγω του συνταγματικού μας πλαισίου λόγω των παραδόσεών μας ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα, στις, ε, στις δημοκρατίες μας. Και το να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο καταχρηστικό, όπως ονομάζεται, εργαλείο, όπως εφαρμόζετε εσείς στην κρυπτογραφία, την κρυπτογράφηση που λέτε ότι είναι το μέσο των κακών, ε, το να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο λέγεται ότι είναι κατάχρηση. Κατάχρηση δηλαδή αν κάποιος περπατάει στο δάσο και μετά σβήσουμε τα ίχνη του. Οι φιλελεύθερες δημοκρατικές μας κοινωνίες μας το έχουν επιβάλει να το ονομάζουμε αυτό κατάχρηση των ελευθεριών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να αφήσουμε αυτές τις κατηγορίες και να ψάξουμε να βρούμε αυτούς που προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους ε, online χρησιμοποιώντας το δίκτυο Tor και όπως είπατε αυτοί το χρησιμοποιούν ε, αυτό το εργαλείο και ίσως να είναι μια μειονότητα από να προσπαθεί φυσικά να προστατευτεί από εξτρεμιστές που προσπαθεί να τους εντοπίσει και να τους βρει στο σπίτι τους. Μπορεί να μην είναι μόνο στην Κίνα, μπορεί να είναι και εδώ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για κάποιους ανθρώπους να έχουν τη δυνατότητα να κρυφτούν ή τουλάχιστον να κρυφτούν στα σπίτια τους ε, ας εστιαστούμε στην ευκαιρία που μας προσφέρει όλο αυτό που προσφέρει στις αστυνομικέ αρχές εφόσον έχουν εύλογες αμφιβολίες, εύλογες υποψίες ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Φυσικά μπορώ να κρυφτώ στο σπίτι μου αλλά αν υπάρχει κάποια υποψία για μένα, τότε οι αστυνομικές αρχές έχουν τον τρόπο, έχουν τα εργαλεία για να μπουν στο σπίτι μου. Να μπουν και να ψάξουν τα πάντα και να με βγάλουν και από το σπίτι. Έχουμε αυτά τα μέσα στο νομικό μας πλαίσιο. Διαφυλάζονται από νομικές διαδικασίες, πρέπει να υπάρχει δικαστής, πρέπει να υπάρχει ένταλμα κτλ. Να κάνω μια έκκληση λοιπόν εδώ, να καθίσουμε κάτω και να δούμε πώς μπορεί κατά περίπτωση να εφαρμοστούν οι νομικές μας διαδικασίες ε, ερευνών κατοίκων, ε, ερευνών στο διαδίκτυο, να δούμε όλες αυτές τις καταστάσεις στην πραγματική ζωή και στο ψηφιακό περιβάλλον. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει κάποια σοβαρή κλιματική δραστηριότητα ε, κάπου διακίνηση ναρκωτικών μπορώ να κάνω παρακολούθηση με βίντεο υπό συνθήκε. Εάν έχω μια φάρμα σερβερ, ένα σερβερ φάρμα που, τακτικά χρησιμοποιούνται από εγκληματίες, μπορώ για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα να παρακολουθώ τι γίνεται εκεί και να παρακολουθώ το ποιο πηγαίνει εκεί. Α εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτέ τι ευκαιρίε χωρίς να εγκαταλείπουμε τις διαδικασίε που έχουμε στη διαθέση μα τώρα. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ε, χρειαζόταν να εξηγήσω λιγάκι τη θέση μου. Ε, κοιτάξτε, πράγματι, μακρηγορήσατε. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε και μια τεράστια συζήτηση σχετικά με το ευρωπαϊκό ε, ψηφιακό θεματολόγιο. Θα έχουμε πράγματι μια συζήτηση σε βάθος για θέματα κρυπτογράφησης. Μόλις ξεκινάει ο Γιώχαν, στην αρχή είναι πάντα δύο, μετά προκαλεί κάπως και εμφανίζονται και άλλοι. Ε, τώρα έχουμε άλλους έξι τουλάχιστον. Η κυρία Βερζιά έχει το λόγο. Oui, euh, merci. Euh, Ευχαριστώ. Ναι, ναι, πολύ ενδιαφέρον τόσο είπε ο συνάδελφος Άλμπρεχτ και συμφωνώ 100% μαζί του. Κύριε, άκουσα το μήνυμα το οποίο στείλατε. Είναι σαφές. Χρειάζεστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να έχετε επιπλέον μέσα στη διάθεσή σας. Και να μην είναι φραγμός στη δραστηριότητά σας η νομοθεσία. Έχουμε όλο ένα και περισσότερο κυβερνό έγκλημα. Οι δε κυβερνό όλο ένα και περισσότερο βοηθούνται από ειδικού Έτσι είναι. Είναι ευφύ οι εγκληματίε, άρα και εμείς θα πρέπει να αποσαρμοστούμε. Αυτά τα θέματα με ενδιαφέρουν από πολλά χρόνια. Γι' αυτό και όντω συνεχώς θέλουμε περισσότερα μέσα να δράσουμε. Λιγότερο να μας δίνει τα χέρια η νομοθεσία και να έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα. Πάρα πολύ σωστά μας το είπατε κύριε. Σταματάμε του εγκληματίες με μεθόδους παραδοσιακές. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τα μέσα ούτως ώστε κανείς να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που υπάρχουν. Δεν είναι μόνο τα μέσα που βοηθάνε. Ε, υπάρχει το πρότυπο το κινέζικο, το ρώσικο. Όχι, όχι, όχι. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε και να προσαρμοστούμε για τα μέσα μας. Να μην καούν τα χολορά μαζί με τα ξερά. Μας είπατε ένα σωρό αριθμητικά στοιχεία το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυτικά. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι το συγκεκριμένο. Γιατί όταν λέμε ότι όλο ένα και πιο νέα είναι τα θύματα κάτω από δύο ετών, μα αν κανείς ενδιαφέρεται τα μαθαίνει. Και το μόνο μέσο να το αποφύγουμε αυτό είναι η πρόληψη, παιδεία όσο πιο νωρίς γίνεται. Δεν πιστεύω ότι η εφαρμοστέα μέθοδος εδώ είναι η πιο σωστή. Δεν έχω πιστεί από αυτά τα επιχειρήματα. Επίσης είπατε ότι η νομοθεσία δεν παρακολούθησε την τεχνολογία, άρα θα πρέπει η οδηγία να μας βοηθήσει. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Τι χρειάζεστε γιατί όλα αυτά τα οποία άκουσα μου δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν κάνουμε τίποτα, γυρίζουμε γύρω γύρω από το ίδιο πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να μπλοκαριζόμαστε από τις αρχές και πεπιθήσεις μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο επόμενος. Να, κάποιες ερωτήσεις, πρόκληση που έχει ο Ρόμπ να απαντήσει. Θα του δώσουμε τώρα το ρόλο για να απαντήσει και θα πρέπει και να συζητήσουμε για το θέμα του κύριου Κέρκοπ για το PNR, τα στοιχεία των επιβατών δηλαδή. Άννα Γκόμες είναι η επομένη. Καταλαβαίνω το σκεπτικό των συναδέλφων Άλμπρεχτ και Βερζιά και επίσης ε, το καταλαβαίνω ακόμα καλύτερα διότι τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια ε, ολιγορία σε σχέση με την ε, εφαρμογή της τάξης όχι απαραίτητα εκ μέρους τους ε, Europol, αλλά εκ μέρους ε, κυρίως ε, υπηρεσιών, ε, μυστικών υπηρεσιών και γι' αυτό τον λόγο φτάνουμε σε αυτήν την επιφυλακτικότητα που υπάρχει χωρίς αμφιβολία. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι εδώ πρόκειται για μία συνέπεια της εξέλιξης της τεχνολογίας και μάλιστα του γεγονότος ε, ότι δεν υπάρχουν οι πόροι τους οποίους ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν την ε, εγκληματικότητα με αυτή την τεχνολογική εξέλιξη. Έχουμε ένα πραγματικό έλλειμμα και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό παντού και για όλους, αλλά εγώ υπήρξα ήδη έγκλημα του κυβερνό χώρου κυρίως όταν έκανα τις έρευνές μου για τη διαφθορά. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά οι αρχές ε, στις οποίες τράφηκα ήταν απόλυτα ε, αδύναμες και ανίκανες ε, να αντιδράσουν, πόσο μάλλον να εντοπίσουν τους υπέτειους. Έτσι λοιπόν θα μπορούσε στη δική μου την περίπτωση να, έχει, να είναι κάτι που να έχει σχέση με την ε, εκμετάλλευση και κακοποίηση των εγγονών μου. Και να σας πω την αλήθεια, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, εγώ θα τασόμουν υπέρ της ε, απώλειας βασικών ελευθεριών για να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα. Και εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για τις βασικές ελευθερίες. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τα νέα μέσα που χρειάζονται οι υπηρεσίες δίωξης εγκλήματος, ε, τα νόμιμα μέσα που χρειάζονται, τις ε, νόμιμες προϋποθέσεις. Και δεν μπορούμε να τα γνωρούμε όλα αυτά. Και αυτή είναι μια ερώτηση προς τον κύριο Ράιτ. Δηλαδή είναι απολύτως απαραίτητο κάπως να τα βρούμε με πολύ σημαντικούς εταίρους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες γιατί ξέρουμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες δεν υπάρχει νομοθεσία για την ιδιωτική σφαίρα και αυτό κατά κάποιον τρόπο μάλιστα υποθάλπει την εγκληματικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο Βεβαίως και οι δικοί τους οι υπάλληλοι ε, των ε, Ηνωμένων Πολιτειών κάνουν, προβαίνουν και αυτοί σε καταχρήσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα. Η Μόνικα Χολμάια έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν τρεις ερωτήσεις. Θέλω να κάνω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά στο εξής. Θα πάρω ένα παράδειγμα. Ε, πιστοτικές κάρτες, απάτη. Κάποιος βλέπει, ας πούμε, ότι στο λογαριασμό του λείπουν 2.000 ε, ευρώ. Συνήθως η τράπεζα το επιστρέφει το ποσό και από τη στιγμή που γίνεται αυτό σταματούν οι αστυνομικές έρευνες. Και ρωτώ στη Europol Πόσες πληροφορίες καταφτάνουν σχετικά με αυτές τις ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις από τα κράτη-μέλη για να μπορεί η Europol να φτιάξει ένα μοντέλο. Γιατί δεν πρόκειται συνήθως για 2.000 ευρώ, πρόκειται για πολλά, πολύ περισσότερα χρήματα, εκατομμύρια ευρώ και μόνο που τα ποσά αυτά επιμερίζονται μέσω του διαδικτύου σε περισσότερους ε, αποδέκτες όχι ας πούμε που συμβαίνει σε μια ληστεία όπου το ποσό που ε, παίρνει κανείς ε, το παίρνει μια φορά και είναι πολύ μεγάλο. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω σχετικά με τις πληροφορίες. Το δεύτερο που θέλω να γνωρίζω είναι το εξής. Ο συνάδελφος Αλμπρέχτ ε, αναφέρθηκε στην διατήρηση των δεδομένων. το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρθηκε σε θέματα αναλογικότητας και από την άλλη είπε ότι ο περιορισμός των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται αποδεκτός όταν πρόκειται για θέματα ασφάλειας των πολιτών. Κατ' ουσίαν εδώ ε, πρόκειται για το εξή. Ε, έχουμε δύο θεμελιώδη δικαιώματα που παλεύουν μεταξύ τους στην οδηγία περί διατήρησης ε, δεδομένων Εκεί αναφέρεται ότι θα πρέπει κανείς ε, να προχωρήσει σε τοπικό επίπεδο, με τοπικές ε, δράσεις, ας πούμε με την παρακολούθηση μέσω βίντεο. Γι' αυτό λοιπόν, μήπως μπορείτε εσείς ε, έτσι κάπως να μας ενημερώσετε για το κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες περιορισμού στον χώρο των υπολογιστών και αν ναι, τι είδους δυνατότητες είναι αυτές και από την άλλη εσείς εξαρτάστε πλήρως από κάποια δεδομένα τα οποία αν δεν τα έχετε στην περίπτωση αυτή ε, είσαστε έρμεα της διεθνούς εγκληματικότητας. Μήπως μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιους δείκτες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και στην πολιτική μας εργασία. Μία τρίτη ερώτηση. Οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι ασχολούνται με το διαδίκτυο και όλες τις ε, τεχνικές μορφές της εγκληματικότητας. Τόσο στη Europol αλλά και στα κράτη-μέλη υπάρχουν, υπάρχει άραγε επαρκές προσωπικό το οποίο να είναι σε θέση ακριβώς ε, να προβλέψει αυτή τη διάσταση του προβλήματος ή μήπως ε, εξακολουθούμε να υποφέρουμε από έλλειψη προσωπικού και στην περίπτωση αυτή η εγκληματίες να είναι σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς. Νίκα, σε ευχαριστούμε. Επόμενος κύριος Πόνη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε για την ε, παρουσίαση. Νομίζω ότι μας δημιουργεί πάρα πολλές ε, προτάσεις ε, και ιδέες ε, με τα συμπεράσματα τα οποία περιέχει η σχετική έκθεση. Επίσης, όταν συζητούμε για την ε, ψηφική παράσταση θα πρέπει να ενθυμούμεθα ότι έχουμε κάποιες νομικές διατάξεις που ισχύουν στον πραγματικό κόσμο. Επίσης θα πρέπει την ε, υλοποίηση των όσων αποφασίζουμε να εφαρμόζουμε τα ίδια και στον ψηφιακό κόσμο και στον πραγματικό κόσμο. Να ε, γίνεται λοιπόν η σχετική προσαρμογή. Εξαπλώνεται το κυβερνό έγκλημα και άρα η κυβερνό ασφάλεια από πάση απόψεω είναι η πρόκληση για όλους μας. Νέα αρχιτεκτονική χρειάζεται για να υπάρχει περισσότερη ισορροπία μεταξύ της προστασίας του ιδιωτικού βίου και της ασφάλειας, της δημόσιας ασφάλειας και της ατομικής. Έχω δύο ερωτήσεις. Δεν είναι μόνο για εσάς ε, κύριε Γουενράιτ, αλλά είναι και για εμάς τους ίδιους. Πρώτα πρώτα, πώς είναι δυνατόν να συγκεράσουμε ε, το, το νομικό πλαίσιο για την προσθέτηση των δεδομένων με κάποιες νέες δυνατότητες που υπάρχουν όσον αφορά την ε, ε, τις λύσεις για την προστασία του ιδιωτικού βίου αλλά και την προστασία της βιομηχανίας. Επίσης, πώς μπορούμε να επανακαθορίσουμε το θέμα της διακράσης των δεδομένων κατόπιν της απόφασης του δικαστηρίου. Πώς θα, θα είναι αυτές οι λύσεις αποδεκτές από τον κόσμο που τους αφορά όσον αφορά τις προσδοκίες τους και πώς όλα αυτά θα είναι πιο χρήσιμα για την αστυνομία της έρευνας κλπ. Χρειάζεται να βρούμε ισορροπία αν θέλουμε να προστατεύσουμε την κοινωνία, τα φυσικά πρόσωπα και ταυτόχρονα λοιπόν να προστατεύσουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γκρίσπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη και ακριβής. Λίγα λόγια για να κάνω δύο ερωτήσεις. όπως έχουμε ε, συνηθίσει εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, να κάνω λοιπόν δύο ερωτήσεις ε, για το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια ισορροπία σε αυτό το τομέα της δημοκρατίας μεταξύ της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και της προσπάθειας να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις δυτικές δημοκρατίες. Αλλά τα νούμερα που αναφέρατε θα αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα. Είναι τρομακτικά τα νούμερα της παιδικής πορνογραφίας που καταδεικνύουν αυτόν τον τεράστιο πολλαπλασιασμό, τη διάδοση, την τρομακτική σοβαρή διάδοση των περιπτώσεων εκμετάλλευσης και βίας κατά ανηλίκων. Φυσικά υποστηρίζουμε τα κέντρα ερευνών, την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, αλλά όπως βλέπετε είναι σαν να ανεβαίνουμε αντίθετα μια κυλιόμενη κλίμα, κλισκάλα. Όταν προσπαθούμε να επιτύχουμε αυτή την ισορροπία, έχω δύο συστάσεις γι' αυτό. Και εσείς είπατε προηγουμένως ότι είμαι άνθρωπος, όχι πολιτικός. Να σας πω ότι και εμείς ζούμε στην πραγματική ζωή, όπως και εσείς. Και η Αναγκομέζη πένθεμισε την εμπειρία της και δικός μας ρόλος είναι και εμείς να είμαστε κοντά στον πολίτη. και όχι να είμαστε θεωρητικοί. Να σας ρωτήσω λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία, τις ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών, ώστε να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση αυτή και να ασκήσουμε την ευθύνη που έχουμε αναλάβει ενώπιον κυρίως των ε, νεότερων σε ηλικία που εξορισμού είναι πιο ευάλωτοι και πρέπει εμείς να προστατεύσουμε με όλα τα μέσα. Και δεύτερον, ε, πώς θα γίνει αυτό σε ένα νομικό πλαίσιο εφάμιλο των ε, ιδεολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά λοιπόν την παιδική πορνογραφία, ίσως θα έπρεπε να φτάσουμε μέχρι το μπλοκάρισμα των ιστοσελίδων. Θα πρέπει να είναι κάτι δυνατό. Αυτό όμως μπορεί να γίνει σωστά μόνο εντός ενός οργανωμένου ευρωπαϊκού πλαισίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Νάταλη. Ο καταλόγος των ομιλητών έχει κλείσει τώρα γιατί έχουμε και το σημείο για το PNR μετά από αυτό. Ακολουθεί η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, άκουσα με πολύ προσοχή. Μήπως κάτι λείπει στην έκθεση αυτή. Όταν μιλάμε για κρατικούς οργανισμούς, που είναι θύματα επιθέσεων. Στο Βέλγιο υπήρξε στόχος ε, hacking το σύστημα της Belgacom, ε, του γίγαντα των τηλεπικοινωνιών, όπως φαίνεται από την Αμερική. Αυτό συνέβη πρόσφατα. Και πιθανότατα να υπήρξαν παρόμοιες επιθέσεις από τη Ρωσία. υπήρξαν επιθέσεις στις χώρες της Βαλτικής. Δεν βλέπουμε να συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές τις επιθέσεις στην έκθεση. Πρόκειται για μια κατάχρηση, για ένα έγκλημα. Μπορεί να μην είναι οργανωμένη η εγκληματικότητα, αλλά είναι έγκλημα το να επιτίθεται μια χώρα στα συστήματα μιας άλλης. Έχετε μελετήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτό. Γίνεται κάποια συζήτηση εσωτερικά για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Και όσον αφορά τους κινδύνους ε, παρίσφρησης από άλλες αρχές, από άλλες κυβερνήσεις, από τη Ρωσία, από την Κίνα. σε ευαίσθητες πληροφορίες. Έχετε κάποια εικόνα αυτού του κινδύνου. Και κάτι δεύτερο για τα θεμελιώδη δικαιώματα συζητήσαμε πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν μιλάτε για την εκμετάλλευση ανηλίκων. Είναι κάτι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει, αλλά δεν μπορούμε να παραιτηθούμε των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όποιος ε, συμπεριφέρεται καλά, πληρώνει την κακή συμπεριφορά άλλων. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο, έναν ενδιάμεσο τρόπο για να καταπολεμήσουμε αυτέ τι περιπτώσει εκμετάλλευση. Το να εγκαταλείψουμε στο σύνολό του τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μου φαίνεται ότι είναι σαν να βλάπτουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να δούμε τις, ε, ε, εταιρείε ε, παροχή υπηρεσιών ίντερνετ όπω η Google και τι εταιρείε που παράγουν ε, υπολογιστέ. σω αυτέ θα μπορούσαν να μα βοηθήσουν στο να αντιμετωπίσουμε την εγκληματικότητα. Ίσως εκεί να υπάρχουν δυνατότητε να μελετήσουμε τι περιπτώσει αυτέ. Ε, χρειαζόμαστε ανθρώπου εκπαιδευμένου στους υπολογιστές, στα λογισμικά, αλλά να είναι εκπαιδευμένοι και στο moral hazard, στους ηθικούς κινδύνους. Δεν μπορεί να είναι κλασικής μορφής ε, συνεργάτες Πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να αντιλαμβάνονται τις περιπτώσεις να καταλαβαίνουν τις ενδείξεις κατάχρησης. Ευχαριστώ. κύριος Ματέρα. Κυρία Ματέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι σύντομη. Και η προηγούμενη συνάδελφος ε, επέστησε την προσοχή στο ίδιο ζήτημα. Θα επαναλάβω τα ίδιο και είναι σημαντικό ο κύριος Διευθυντής να απαντήσει στην, αυτή, στην ερώτηση αυτή. Μιλάμε για εφαρμογή μέτρων υπεράσπισης των νέων χωρίς να πλήξουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό και μετά εσείς μιλήσατε για μια συνεργασία μεταξύ οργανισμών. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν συνεργασία, με, ε, δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ΣΕΠΟΛ και Ευρωπόλ. Ευχαριστούμε που τηρήσατε το χρόνο. Πρόεδρος η Μπέργκη τελευταία. Και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Και εγώ θα είμαι σύντομη όσον αφορά την εμπλοκή των ε, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή του νόμου. Και το ερώτημα είναι όχι το αν θα το κάνουμε ή όχι, αλλά σε ποιο βαθμό. Γιατί οι ιδιώτες δεν μπορούν να αναλάβουν την εφαρμογή του νόμου να συλλάβουν κάποιον αλλά εάν έχουν υπόψη τους ότι θα γίνει ένα έγκλημα να ενημερώνουν την ε, αστυνομία. Άρα να δούμε μέχρι ποιο σημείο οι επιχειρήσεις ε, είναι εδώ να συνεργαστούν με την αστυνομία. Και πού θα είναι η κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να περιβεί κανείς τώρα όσον αφορά το άλλο θέμα, την ε, χρησιμοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την εφαρμογή του νόμου. Εδώ πέρα υπάρχει κάποιο όριο γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Όποτε έχουμε να κάνουμε με τέτοια φορτισμένα ζητήματα όπως η σεξουαλική κακομεταχείριση των ανηλίκων, πάντοτε είμαστε πιο πρόθυμοι να πούμε εντάξει, θα πρέπει να περιστύλουμε τα δικαιώματα γιατί είναι κάτι που πλήσει τα παιδιά. Αλλά τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε δεν θα αφορούν μόνο την κακοποίηση των ανηλίκων. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει πραγματικά να συζητηθεί είναι το τι θα γίνει με τους κανόνες που έχουν να κάνουν με την πραγματική ζωή και τι κανόνες θα έχουμε στην διαδικτυακή ζωή γιατί είναι θέμα να προστατεύσουμε τα παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της κομμεταχείριση των ε, γυναικών, αλλά γιατί ακόμα και για τους ανηλίκους συνήθως το έγκλημα γίνεται ε, μέσα στο σπίτι. Τι να κάνουμε, ο, ο Γιάννη μας το πελίγο λαϊκίστηκα ότι μπορούμε να βάλουμε ε, σε κάθε σπίτι μέσα μία κάμερα. Βεβαίω και δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Άρα ποια είναι η λύση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο φορτισμένοι και να αντιδρούμε εν θερμό, αλλά χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση για το τι θα κάνουμε, πού είναι το όριο μεταξύ καταπολέμησης εγκλήματος και προστασίας των ελευθεριών και σε ποιο βαθμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή πληροφορία, ποιο μπορεί να έχει πρόσβαση. Το όλα αυτά τα θέματα πρέπει να ζητηθούν και νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε επί τη βάση πραγματικών περιστατικών και όχι συναισθημάτων. Μπρίξ, ευχαριστώ. Και τώρα για να δούμε, ε, όπως κανείς μπορούσε να προβλέψει μεγάλο τον ενδιαφέρον και άρα πολλοί οι ομιλητές. Ρομπ, έχουμε μια έκθεση της πρωτοβουλίας, έχουμε τριμερή διάλογο και άρα θα επανέλθεις. Άρα εάν δεν έχεις το χρόνο να τα καλύψεις όλα σήμερα, οι συνάδελφοι θα πρέπει να ξέρουν ότι θα επανέλθεις συντόμως. Κάνε λοιπόν ό,τι μπορεί για να απαντήσει όσο μπορεί περισσότερα. Ευχαριστώ και πάλι Πρόεδρε. Βεβαίω και συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούσαμε τελευταία ομιλήτρια ότι δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε σε συναισθήματα αλλά σε πραγματικά περιστατικά και στοιχεία. Ειλικρινά, δεν ξέρω αν όλοι καταλαβαίνετε την φύση του προβλήματος. Εάν θεωρείτε ότι μόνο η πρόληψη στον πραγματικό κόσμο και ότι μόνο η τοπική αστυνομία κάτι πρέπει να κάνει στα σπίτια και αυτό θα αρκεί για να σταματήσει να υπάρχει το πρόβλημα σε επίπεδο Ιντερνετ. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη πρόληψη. Βεβαίω θα πρέπει να κάνει περισσότερη αστυνομία, να αστυνομεύσει τα σπίτια εκεί όπου γίνονται όλα αυτά. Γιατί βέβαια πρέπει να σα πω ότι κάθε τοπική αστυνομία έχει μια μονάδα που αφορά ε, ε, Τέτοιου εγκληματίε. Ε, το αυτό τι σημαίνει όμω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα σε επίπεδο ίντερνετ γιατί έχουμε 4 εκατομμύρια ε, συνέχεια που ανεβαίνουν στο ίντερνετ. Το είδαμε με μόνο μία επιχείρηση το είδαμε αυτό. Κύριε Βερσιάρ πρέπει να σα πω ότι ε, θεωρώ βασικό να παληθεύουμε τα στοιχεία μας και δεν, δεν είναι επιφανειακό αυτό που για τα θύματα κάτω από δύο έτη. Ε, το 20% όλων των φόρουμ, μιλάμε 2,5 εκατομμύρια χρήστες που, που μας, μας αφορούν. Και είναι ανεξάρτητη αυτή η έρευνα. Το 20% λοιπόν αυτών των φόρουμ αφορούν μόνο ε, κακομεταχείριση ανηλίκων. Να η πραγματικότητα. Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε και στον πραγματικό κόσμο και στο ίντερνετ. Και εγώ σας λέω να υπάρχει αναλογία. Αναλογία ε, ισχύω και δυνατοτήτων, όχι χωρίς να καταπατούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, να υπάρχει ισορροπία. Υπάρχει ευαισθησία και να μπορούμε να έχουμε απόρριτο τραπεζικό, να μπορούμε να έχουμε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνδιάλαξη, όλα αυτά σημαντικά. Αλλά θα πρέπει και η αστυνομία να έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα τραπεζικά στοιχεία, να, τα, τα, φορολογικά στοιχεία, τους λογαριασμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τέτοια τεχνολογία που είναι φραγμός στην αστυνομία ούτως ώστε να μπορεί να, να, να βρει τους εγκληματίες λόγω της, ε, της κρυπτογράφησης. Αυτό είναι το αδύνατο σημείο επίσης. Ότι δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες στο Ιντερνετ όπως έχουμε στον πραγματικό κόσμο. Και δεν υπερβάλλω. Σας διαβεβαιώ ότι αυτά όλα τα διαπιστώνουμε κάθε μέρα. Έχουμε τώρα πολλές ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις. Χολμάιερ, Γκόμες, πολύ σημαντικές ερωτήσεις για τα κρατημέλη ε, όπου έχουμε όντως εμπλοκή πολύ σοβαρή των ε, κρατών μελών. Δεν παραπονιέμαι ότι δεν μας δίνουν αρκετές πληροφορίες, απλώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τα κρατημέλη έχουν εμπλακεί περισσότερο στην κατάσταση του κυβερνοεγκλήματος παρά αλλού. Το λέω και το ξαναλέω, το κυβερνητικό τα ακούτε, ξέρω, αλλά θέλουμε περισσότερη προοικοδότηση. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά και με την αποκρυπτογράφηση, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό πιέζει περισσότερο από όλα. Τέλος, γιατί η κυρία Βερζιά, μεταξύ άλλων, ε, μας είπε τι ζητάμε. Σας είπα ξεκάθαρα στην εισήγησή μου. Θέλουμε να έχουμε και για το κυβερνέγκλημα τα ίδια μέσα, όπως και τον πραγματικό κόσμο. Να μπορούν οι ιδιωτικέ αρχέ να ανταλλάξουν στοιχεία. Και ο σχετικό κανονισμό να μα δίνει τη δυνατότητα να αναζητούμε πληροφορίε από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα πρέπει αυτό να βγει από την πρόταση του κανονισμού. Και η καταγράφηση, η διακράτηση δεδομένων τέλο πάντων χρειάζεται για να δούμε πώς θα υπερκεράσουμε το μεγάλο μας πρόβλημα την αποκρυπτογράφηση πρόθυμα θα ξανέλθω να σας δω. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε. Ο Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Είχαμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι πολύ σωστά διακρίνεται τις πιο ζουμερές ε, ε, ερωτήσεις να απαντήσετε, θα επανέλθετε. Ευχαριστούμε και μας βοηθήσατε για δύο θέματα μέσα στις διάταξεις Σας παρακαλώ σε αυτό που είπε ο κύριος Άλμπερτ στην αρχή για το έργο της ε, Europol. Να τα ακούνε ιδίως οι νεότεροι εδώ. Συνάδελφοι, τώρα θα πάμε στο σημείο της διάταξης για τα δεδομένα των επιβατών. Um, um, όπως θα θυμάστε συναδελφοί και αυτό φορά κυρίως τους συναδέλφους που τώρα βλέπουν αυτό το ζήτημα. Ο συγητής μας είναι εδώ ο κ. Κέρκο. Σκιώδης ε, είναι ε, κύριος Βος, Ιαν Αλμπρέχτ, Κονίρια Χέρστ και Λάουρα Φεράρα. Θα σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή ειδικότερα για τα νεότερα μέλη. Μια μικρή σύνοψη. Όπως θα θυμούνται οι συναδελφοί, το ζήτημα συζητήθηκε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ κατά την τελευταία θητεία εκείνη την εποχή. Συζητήθηκαν τα ακόλουθα η αναγκαιότητα της πρότασης, το αντικείμενο όσον αφορά τα εγκλήματα όσον αφορά τις ε, εγχώριες ε, και εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης πτήσης, ε, κεντρικό ή αποκεντρωμένο σύστημα, υποχρεωτικό ή καθεξής. Και εκείνη την εποχή η πρόταση απορρίφθηκε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τον Απρίλιο του 2013 με την επακόλουθη πρόταση στην Ολομέλεια να αναπαινθεί το ζήτημα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολλά μέλη έχουν ήδη εισάγει ένα τέτοιο σύστημα ή συμμετέχουν σε πιλωτικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Επιτροπή. Μετά από την απόφαση για τη διατήρηση δεδομένων του δικαστηρίου, τέθηκε το ζήτημα των συνεπειών από μια τέτοια απόφαση. Όπως θα θυμούνται οι συνάδελφοι, αναφέρθηκε από τον Επίτροπο Αβραμόπουλο επίση το ζήτημα. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη έθιξαν το ζήτημα σε σχέση με τους ξένους μαχητές. Σήμερα θα κάνουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. Θα εξετάσουμε πρώτα τα όσα έχει να μας πει ο κύριος Συγητής, ο κύριος Κέρκοπ, μετά το Συμβούλιο, μετά νομίζω η Επιτροπή και θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ των μελών. Τίμωθη λοιπόν σας δίνω το λόγο. Ξεκινήσω εγώ. Uh, ε, θα ήθελα να σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μας προσφέρεται η ευκαιρία να συζητήσουμε για την οδηγία περί των PNR δεδομένων και που θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όπως είπατε πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή αυτή απέριψε την οδηγία Μικρή βέβαια διαφορά και η Ολομέλεια αποφάσισε ότι η Επιτροπή πρέπει να το ξαναδεί το θέμα για να προχωρήσουμε. Σε προηγούμενες ε, περιπτώσεις ε, είχαμε συμφωνίες οι οποίες αρχικά είχαν ε, απορριφθεί σε επίπεδο επιτροπής μετά όμως προχώρησαν αυτές οι συμφωνίες και κατέληξαν μετά από δουλειά σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Βεβαίως τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον συνεργαστούν όλοι και υπάρχει και καλή και υπάρχει και σχετική βούληση. Το Κοινοβούλιο προσκάλεσε πολλούς εμπειρογνώμονες από τον τομέα της ασφάλειας για να μιλήσουν στην Επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια και έχουμε παράδειγμα σήμερα αλλά και άλλες φορές. Και ο κατάλογος όπως γνωρίζετε ε, περιλαμβάνει όχι μόνο τον κύριο Wainwright που ήταν σήμερα και τον κύριο Ζεκέτρο που ήταν συντονιστή ε, περί αντιμοκρατία. Είχαμε εκπροσώπους του Συμβουλίου Ζαν Πολ Λαμπόρντ, ε, ειδικό για αντιτρομοκρατία των Ηνωμένων Εθνών και βεβαίω ε, είχαμε και την κυρία Σεσίλε Μάρστρομ, την ε, πρώην αρμόδια επίτροπο για αυτό το θέμα για ένα αρκετά μεγάλο ε, χρονικό διάστημα και νομίζω ότι τώρα έχουν περάσει περίπου δυόμιση χρόνια από τότε που ξεκίνησα και εγώ να ασχολούμαι με το θέμα. Όλοι λοιπόν όσοι ήρθαν εδώ ε, επισήμαναν ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρξει ένα σύστημα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους φακέλους επιβατών για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και αυτό είναι απαραίτητο για να αντιμετωπιστούν τα αίτια της ε, τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι εργαλείο ε, που πρέπει να χρησιμοποιεί κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διώκονται ορισμένα πολύ σοβαρά εγκλήματα που αντιμετωπίζουμε. Οι φάκελοι των επιβατών αποδείχτηκαν καθοριστικής σημασίας ε, ε, για τους ε, πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγαίνουν στη Συρία, ε, στο Ιράκ, εκεί πηγαίνουν να αγωνιστούν και μετά να επιστρέψουν ε, πίσω στην Ευρώπη. Με το φακέλους αυτούς ε, μπορούμε να εντοπίσουμε τη διαδρομή τους και να εμποδίσουμε αυτούς και άλλους να επιτύχουν τον στόχο τους, τον κακό τους σκοπό. Επίσης βοήθησαν οι φάκελοι στο να ε, συλληφθούν εκείνοι οι οποίοι προβάλλουν ε, άσεμνες εικόνες ε, παιδιών. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες ανησυχίες, το ακούσατε αυτό σήμερα το πρωί και είναι πραγματικά ιδιαίτερα τρομακτικό το να υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα PNR για να εντοπίσουν την ε, διακίνηση ναρκωτικών από την Καραβική στην Ευρώπη. 14 μέλη του οργανωμένου εγκλήματος ε, ε, καταδικάστηκαν συνολικά μέχρι και 79 χρόνια φυλακή. Επίσης τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη διακίνηση γυναικών στην Ιγυρία αλλά και σεξουαλική εκμετάλλευση στη Γαλλία. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό υπόπτων και κάποιους συγκεκριμένους λογαριασμούς και μεθόδους πληρωμής. Με τον τρόπο αυτό ε, θα προέκυπταν πολλά νέα θύματα. Αυτές είναι ενδεικτικά κάποιες ε, περιπτώσεις. Δεν θέλετε να αναφέρω κι άλλες γιατί θέλω να είμαι σύντομος. Ε, Μη ενδεικτική ενδεικτικά, όπως σας είπα, ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις και ένα παράδειγμα για τα θέματα τα οποία εξετάζουν καθημερινά οι υπηρεσίες δίωξη εγκλήματος. Θέλω να καταστήσω σαφές, δεν ήρθα εδώ σήμερα για να πω ότι το PNR είναι το καλύτερο όπλο για την αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να προστατεύσουμε τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων για τους οποίους φέρουμε ευθύνη, δηλαδή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά μόνο τις υπηρεσίες δίωξης εγκλήματος που αυτό πρέπει να το υιοθετήσουν ως πρώτη προτεραιότητα. Για χρόνια ολόκληρα η ε, ε, βιομηχανία, ο κλάδος των ε, αεροσκαφών έχει επισημάνει το πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσουμε στον τομέα και να υπάρχει σχετική οδηγία. Επειδή όμως δεν υπάρχει, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν να κάνουν με 28 διαφορετικά συστήματα τα οποία πολλές φορές προέρχονται μάλλον και διαφορετικά συστήματα από το ίδιο κράτος μέλος. Αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό το σύστημα και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι η προστασία των δεδομένων των επιβατών ποικίλει κατά πολύ ανάλογα ε, με το κράτος μέλος. Συνάδελφοι, μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή οι αεροπορικές εταιρείες ε, αντιμετωπίζουν αιτήματα για πάνω από 50 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα περιεκτικό πλαίσιο και αυτό θα ήταν το πρώτο βήμα για να υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε αιτήματα για μεταβίβαση στοιχείων επιβατών αλλά και για την αρμοδιότητα των ε, υπηρεσιών να πούνε όχι όταν πρόκειται για στοιχεία επιβατών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ε, αν μεταβαστούν υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Υπάρχουν λοιπόν εδώ αρκετοί που έχουν άμεση εμπειρία της τρομοκρατίας, ξέρουν τι σημαίνει και κατανοώ λοιπόν ότι αυτό το θέμα δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Ξέρω ότι έρχονται κάποιοι από χώρες ε, όπου υπάρχει πρόβλημα με τις ελευθερίες, αλλά εκεί ε, υπάρχει και πρόβλημα τρομοκρατίας. Δεν θέλω να μειώσω ε, τη σημασία όλων αυτών που λέγονται για την προστασία των δεδομένων, αλλά ξέρετε αυτή τη στιγμή 15 κρατημέλη έχουν χρηματοδότηση από την ε, Επιτροπή ε, οικοδομούν συστήματα PNR, Λετβία, Εστονία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Λιτουανία και βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και κάποιες άλλες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τους δικούς μας τους κανόνες, ε, τις δικές μας ε, τις ε, προδιαγραφές για όλα αυτά τα συστήματα PNR, γιατί με τον τρόπο αυτό θα καλύψουμε ένα σημαντικό κενό και πρέπει να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε χάος και περισσότερα προβλήματα. Βεβαίως πολλοί λένε ας περιμένουμε ε, μέχρι να υπάρχουν νέοι αρμόδιοι για τη διατήρηση των δεδομένων και για την προστασία τους. Όμως αυτό θα μπορούσε να, να ε, χρειαστεί πολύ χρόνο οι πληροφορίες θα συνεχίσουν να ανταλλάσσονται χωρίς όμως ένα σωστό ε, πλαίσιο και γι' αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες δίωξης. Ως νομοθέτες δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό, κυρίως ε, ε, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι επιχείρημα απέναντι σε μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες διατήρηση δεδομένων θα ισχύουν ε, για αυτή την οδηγία μόλις εγκριθεί η σχετική οδηγία. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραμμίσω στους βουλευτές ότι εγώ πραγματικά επιθυμώ να υπάρξει συμβαστική πρόταση. Μια οδηγία που θα ε, είναι ικανοποιημένη όλοι, η δική μου πόρτα είναι πάντα ανοιχτή, αυτό το γνωρίζουν οι συνάδελφοι από το παρελθόν, Όποιο θέλει να έρθει για να συζητήσουμε επιφυλάξεις του, και εκτός αυτής της Επιτροπής είναι ευπρόζεκτος. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούμε να διώξουμε τους εγκληματίες. Οφείλουμε λοιπόν να αναζητήσουμε μια λογική εξέλιξη του θέματος η οποία βέβαια να επιτρέπει και τη δυνατότητα να προχωράμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ Τίμωθη ε, δεν έχει βάλει βουτυκνό το πόδι στο νερό, αλλά όλο στο σώμα. Να δώσουμε το λόγο τώρα στο Συμβούλιο. Έχουμε δύο συναδέλφους από ό,τι μου έχουν επισημαίνει. Πρέπει να μιλήσετε και οι δύο. Εδώ πρέπει να μιλήσει μόνο ένα σας. Έχουμε χρόνο μόνο για έναν ομιλητή. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο Φιλίππο Κολόμπο, μιλώ εξ ονόματι του Συμβουλίου. Λέγομαι Φιλίππο Κολόμπο από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα εξ ονόματος της Προεδρίας την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί την πρόταση αυτή που μας αφορά ιδιαίτερα. Όπως η κυρία Πρόεδρε, το Συμβούλιο Έχει ήδη καταλήξει συμφωνία το 2012 για αυτή την πρόταση και ακόμα πρόσφατα σε πολιτικό επίπεδο επαναλάβαμε τη σπουδαιότητα που θεωρούμε ότι έχει αυτό το σημαντικό μέσο. Να υπενθυμίσω ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ης Αυγούστου του 2014 όπου ζητήθηκε από όλους τους συνομοθέτες να συνεργαστούν για να καταλήξουν συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους και να επιθυμήσω φυσικά και όλη τη δουλειά που έγινε πρόσφατα και στο πλαίσιο της συζήτησης για τους ξένους μαχητές, τους foreign fighters, όπως υπενθυμιστεί και εσείς. Εμείς θεωρούμε, όπως είπε ο κύριος συζητητής, ο κύριος Κερχόπ, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο καταπολέμησης σοβαρών περιπτώσεων εγκληματικότητας και τρομοκρατίας. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με τους νομοθέτες ώστε να καταλήξουμε γρήγορα σε κάποια συμφωνία η οποία θα μας επιτρέψει να υιοθετήσουμε το μέσο αυτό. Όλες μας οι αστυνομικέ δυνάμεις επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα του θα μπορούσε να έχει αυτό το μέσο και, και θα μπορούσε να βελτιώσει τα αποτελέσματα στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Έχουμε συνείδηση των ανησυχιών πολλών μελών αυτής της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου γενικότερα και που αφορούν οι ανησυχίες αυτές τα δικαιώματα ε, του ιδιωτικού βίου. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να εργαστούμε ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία η οποία θα επιτρέψει να διασκεδάσουμε αυτές τις ανησυχίες και να καταλήξουμε γρήγορα σε μια κοινή λύση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο στην Κομισιόν. Να αναφέρω ότι έχουμε καλέσει τον ε, κύριο Αβραμόπουλο, τον Επίτροπο, στις 13 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή για να συζητήσουμε το ζήτημα PNR μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα που θα μας παρουσιάσει. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βικτόρια Ανίτση, Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα αξιότιμα μέλη, καλημέρα κύριε και κύριοι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία στην Κομισιόν να πει δύο λόγια για αυτό το σημαντικό θέμα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η συζήτηση για αυτό το θέμα συνεχίζεται. Έχει επανεκκινηθεί σε αυτή την Επιτροπή. Εκ μέρους της Κομισιόν εμείς εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τη λογική στην οποία βασίζεται η πρόταση PNR και η οποία υποβληθήκε το 2011. Υποστηρίζουμε τις ιδέες που οδήγησαν σε αυτό το σχέδιο νομοθετήματος. Δεδομένων αυτών και όπως αναγνώρισε ο ίδιος ο Επιτρόπος ο κ. Αβραμόπουλος στην ακρόασή του ενώπιον της παρουσίας Επιτροπής είναι σαφές ότι η προκειμένη πρόταση πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά με γνώμονα τις αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται στην απόφαση του δικαστηρίου για την οδηγία διατήρησης δεδομένων. Πρέπει επίσης να εξεταστεί με, βάση, με γνώμονα τις κατευθύνες γραμμές του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την αναλογική χρήση των δεδομένων PNR. Εμείς πιστεύουμε ότι η οδηγία πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και πρέπει να φροντίσουμε ότι θα μπορεί να περάσει από οποιαδήποτε αμφισβήτηση του δικαστηρίου. Συνέπω, κύριε Πρόεδρε, η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεργαστεί με του νομοθέτες ώστε να τους προσφέρει αρρωγή για τη διαμόρφωση μιας πρότασης που θα εφεργαμίζεται πλήρως με τις απαιτήσει που προκύπτουν από την απόφαση που ανέφερα και ειδικότερα για να διασφαλίσει την αναλογικότητα των προβλεπόμενων μέτρων όσον αφορά την προστασία των ατομικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίε της Κομισιόν εξετάζουν την πρόταση σε αντιπαραβολή με τα στοιχεία που μόλις ανέφερα. Οι εσωτερικές διαβουλεύσεις ε, λαμβάνουν αυτή τη στιγμή η χώρα εντός της Κομισιόν ώστε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο επιτεύξης αυτού του στόχου αναλογικότητας. Όπως είπατε και εσείς ο ίδιος κύριε Πρόεδρε, ο Επιτρόπος ο κ θα συμμετάσχει στην σύνοδο της Λίμπες της 3 ε, Δεκεμβρίου και με την ευκαιρία θα σας παρουσιάσει συγκεκριμένες ιδέες για το μέλλον. Ευχαριστώ. Okay, thank you. I'm um, Ευχαριστώ πολύ. Να στραφώ τώρα στους Κιώδης με τη σειρά με την οποία αναφέρονται. Ένα Κιώδης δεν ε, ανέφερε ότι θέλει να μιλήσει. Άξελ, είστε τελευταίος. Μπρίγκιτ, παρακαλώ σε επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Για σήμερα να περιοριστώ σε κάποιες γενικού χαρακτήρα παρατηρήσεις για κάποια ζητήματα τα οποία ε, σχετίζονται και με τις ρυθμίσεις που αφορούν τα στοιχεία των επιβατών και σχετικά με αν θυμάστε, τη συζητήσαμε σήμερα το πρωί αλλά και την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Wainwright από την Europol. Ακούσαμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ούτως υπήν όσον αφορά την ροή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών ε, αλλά και μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών και οργάνων. Είπαμε την πρώτη εβδομάδα ότι δεν αξιοποιούμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε για να κατοπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα ε, δεν το κάνουν όλα τα κρατημέλη μελη Επομένως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι τα υπάρχοντα μέτρα αξιοποιούνται γιατί μόνο τότε μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν χρειάζονται και άλλα μέσα και αν μπορούν να μας δώσουν εκείνα προσθέμενη αξία για την καταπολέμηση του εγκλήματος. Δεύτερο, από τότε είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά την διακράτηση των ε, δεδομένων και την σχετική οδηγία. Δεν είμαι νομικός, αλλά κάπως έχω θυμώσει, διότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία πλέον δεν υπάρχει, διότι το δικαστήριο είπε ότι δεν συνάδει προς το κοινοτικό δίκαιο και τις ε, κοινοτικές ε, αξίες. Όμως έχουμε τις οδηγίες των κρατών μελών που μοιάζουν πάρα πολύ και οι οποίες ακόμα βρίσκονται ενισχύει παρά το ότι συμφώνησε όποιος προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ίδιες αξίες και κανόνες δικαίου. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι νομικός. Αλλά για μένα η κατάσταση μου φέρνει μηχανία, έκανε βρισμό, θυμό. Είπε ο κ. Κέρκο, πάρα πολλά κράτη-μέλη παίρνουν τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να χτίσουν ένα τέτοιο σύστημα ε, για τα δεδομένα των επιβατών. Αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές αυτές οι αξίες. Και δεν μιλώ για τις συνέπειες μόνο του δικαστηρίου. Θα πρέπει φυσικά να συμμορφωθούμε. Και επίσης θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό η απόφαση του δικαστηρίου έχει κάποιες επιπτώσεις στα στοιχεία των επιβατών, αλλά και στα άλλα μέτρα τα οποία θα ληφθούν στο μέλλον. Άρα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τώρα το ότι θα έχουμε νέα οδηγία για δεκάτηση δεδομένων και μιλώ για οδηγία. Ο Τίμωθη και είπε ότι ε, μπορεί να περιμένουμε πολύ χρόνο. Συμπαθάτε με αλλά δεν φταίει για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς συζητήσαμε επί μακρόν και τελικά αποφασίσαμε. Παρά το ότι είχαμε ε, επιμέρους διαφορετικές απόψεις από την αρχή της συζήτησης. Τα κράτη-μέλη έχουν βάλει τροχοπέδι στην διαδικασία λήψη αυτής της απόφασης. Άρα εάν θέλουν να λάβουν ε, νέα μέτρα ε, θα, για τη συλλογή των δεδομένων, τότε θα πρέπει να πάνε να βρουν κάποια κοινά στάνταρ, κοινά πρότυπα και ιδίω όσον αφορά την οδηγία. Να ακούσατε τι είπαμε σήμερα, τι είπε και την εβδομάδα ο Ρόμπερτ Βέινράιτ. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι οι κοινέ διατάξει θα πρέπει να καλυφθούν και από την οδηγία και από τον κανονισμό. Και αυτό δεν θα είναι ένα βάρος. Θα είναι, είναι αναγκαίο να υπάρχει κάτι τέτοιο και να έχουμε έτσι αμοιβαία αποδοχή και όσον αφορά την εφαρμογή του, του νόμου και όσον αφορά την δικαστική συνεργασία. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε και να βρούμε επιπλέον μέτρα. Άρα απόκειται στα κράτη-μέλη αν θέλουν να υπάρξει ταχεία μια απόφαση να κάνουν πρώτα-πρώτα αυτό που τους αναλογεί. Αυτά κάπως γενικόλογα που θέλω να πω για το θέμα τώρα. Γιάννη, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επίσης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που μας ενημέρωσε για τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι λυπούμαστε πάρα πολύ που δεν έχουμε την EDPS ε, να παρουσιάσουν και αυτή την άποψή τους ε, μετά την απόφαση που λήφθη σχετικά με την προτινόμενη νομοθεσία. Αυτό θα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ίσως στην επόμενη φάση μπορούμε να το προβλέψουμε. Τώρα, κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι κανείς ε, δεν αντιτίθεται στο να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις υπηρεσίες ε, εφαρμογής του νόμου. Τούν αντίον όλες οι ομάδες ε, συμφώνησαν να υπάρχει ένα ε, ευρωπαϊκό σύστημα ερευνών να μπορούν να ανταλλάσσουμε σε αυτό πληροφορίες οι υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου. Εμείς ασκούμε πίεση γι' αυτό και ειδικά εγώ έχω πιέσει και πολύ ουσιαστικά αν θέλετε, γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι Πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτό δεν λειτουργεί και όλα τα παραδείγματα που μου παρουσιάστηκαν έχουν σχέση με το ότι δεν μεταφέρθηκαν οι πληροφορίες ε, ανάμεσα στις διάφορες αρχές που υπήρχαν. Υπήρχαν για να ε, προληφθεί και να καταπολεμηθεί το διεθνές έγκλημα και οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Η προτινόμενη λοιπόν οδηγία δεν αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών αλλά αφορά στην διατήρηση πληροφοριών. Και εδώ το δικαστήριο αποφάντηκε πάνω σε αυτή την οδηγία και χαίρομαι που η Κομισιόν αναγνωρίζει και το έλεγε αυτό επίσης και ο Επίτροπος, κύριος Αβραμόπουλος, ότι προφανώς θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την προσέγγιση σχετικά με τη συγκέντρωση ενδομένων για τους φακέλους των επιβατών, το PNR. Να δούμε πού μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε. Και θέλω να πω ότι μια βασική διάταξη της απόφασης ε, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Είναι η υπαριθμόν 59 και παραθέτω Επιπλέον, ενώ πρέπει να συνεισφέρουμε στον αγώνα κατά σοβαρού εγκλήματος, η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων δεν απαιτεί να υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δεδομένα τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και την απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Και πιο συγκεκριμένα να μην υπάρχει διατήρηση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή για μια συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη και για συγκεκριμένα άτομα τα οποία κατά τον ΑΒ τρόπο εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα ή δεύτερη επιλογή σε άτομα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να εντοπιστούν σοβαρά εγκλήματα. Τέλος παράθεση. Αυτό λοιπόν είναι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που λέει ότι η διατήρηση δεδομένων πρέπει να ισχύει και για το PNR, αλλά αυτό δεν προβλέπεται στο PNR ούτε χρονικά, ούτε όσον αφορά τη γραφική ζώνη, ούτε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Προβλέπεται η διατήρηση απλά όλων των στοιχείων όλων των ταξιδιωτών που μπαίνουν και βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλετε, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου, όλων εκείνων που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αεροπλάνα. Και αυτό μόνο για πέντε χρόνια. Μετά λοιπόν από αυτή την απόφαση δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και από ό,τι ακούω και η Κομισιόν ε, συμφωνεί ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ λοιπόν προτείνω ότι εφόσον η Κομισιόν βλέπει ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να αναξιολογήσουν την κατάσταση και όχι απλά να προχωρήσουν με μια οδηγία που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που προτείνονται. Και εν πάση περιπτώσει Υπάρχουν ερωτήσεις προς την νομική υπηρεσία σχετικά με αυτή την απόφαση του Απριλίου, άρα θα πρέπει να περιμένουμε αυτούς και να μας ε, παρουσιάσουν τη γνώμη τους κατά πόσον υπάρχει περιθώριο ελιγμών για την εκπόνηση κανονισμών σχετικά με τη διατήρηση δομένων Παραλαμβάνω, εγώ δεν είμαι αντίθετος, είμαι μάλιστα σαφώς υπέρ του να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών και μάλιστα αυτό ή δυνατόν να εφαρμοστεί ακόμα και σήμερα. Και δεν είμαι αντίθετος, σας το λέω η επιπρόσθετη υποχρεωτική διατήρηση που προβλέπεται σε αυτήν την οδηγία αυτό είναι το πρόβλημα και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αγνώντας την απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Next. Ωραία. Στη συνέχεια δίνω αρκετό χρόνο στους σκιώδεις γιατί αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο παραχωρητικός, αλλά τι μου θα έχετε την ευκαιρία και στο τέλος να έχετε αρκετό χρόνο. Ακολουθεί η Κορνήλια, σκιώδης εκ μέρους της Γκουε. Λοιπόν, ε, εδώ δεν σημειώνουμε πρόοδο. Γυρίζουμε γύρω-γύρω από τα ίδια συζητάμε σε όλες τις συνεδριάσεις μας για τους φακέλους επιβατών και καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι η διατήρηση δεδομένων όπως προβλέπεται τώρα στην οδηγία αυτή η διατήρηση δεν είναι συμβατή με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει καμία απολύτως αξία. Νομίζω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως ε, λειτουργούμε τώρα και θέλω να σας επισημάνω ότι ε, το άρθρο 29 λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι σε επίπεδο περιεχομένου δεν υπάρχει κάποια βάση για το PNR στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορίζουν κάποια κριτήρια με βάση τα οποία μπορούν να διατηρούνται μόνο κάποια στοιχεία, όχι γενικά όλα τα στοιχεία για έναν επιβάτη. Και είπαν πρώτον θα πρέπει να ε, διαφυλάσσεται η χάρτα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, να μην παραβιάζεται. Δεύτερον, ε, ειδικέ περιπτώσεις και τρίτον η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών. Υπήρξε λοιπόν η ομάδα εργασία του άρθρου 29 που τα είπε όλα αυτά με απόλυτη σαφήνεια και σε πρόσφατο έγγραφο που εγκρίθηκε εκεί υπάρχει σαφής επισήμανση ότι η αναλογικότητα των μέτρων θα πρέπει να ελέγχεται τόσο των μέτρων που ήδη υφίστανται όσο και άλλων που πρέπει να ληφθούν πριν μάλιστα καν σχεδιαστούν. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Υπήρξε περίπτωση σοβαρής αξιολόγησης ή μιας κάποιας αξιολόγησης για το πώς εφαρμόζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και εάν ναι, αν έχει γίνει αυτή η αξιολόγηση θα ήθελα να γνωρίζω Κομισιόν και Συμβούλιο ποια μέτρα δεν απέδωσαν. Πού βρίσκεται το κενό. Ποια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι απαραίτητο να ληφθούν νέα μέτρα. Και το δεύτερο που θέλω να γνωρίζω από εσάς είναι το εξής τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ε, δείξτε τα μας ε, μπορούμε άραγε να τα αποκτήσουμε ή μήπως δεν έχετε κάνει καθόλου αξιολόγηση. Θα ήθελα οπωσδήποτε να μου τα απαντήσουν αυτά το Συμβούλιο και η Κομισιόν πριν προχωρήσουμε και αναφέρεται συνεχώς ε, το επιχείρημα ότι στα κράτη-μέλη θα ε, συνταχθούν συστήματα PNR, γι' αυτό πρέπει να εναρμονιστούμε. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε το λάθος να διαθέσει χρήματα για αυτό το σύστημα. 50 εκατομμύρια εκατομμύρια. Έδωσε 50 εκατομμύρια χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη βάση. Διοχετεύονται χιλιάδες ε, εκατομμύρια στα κράτη-μέλη και μετά το ερώτημα πώς μπορεί να προκύψει ένα ενιαίο σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια ψευτοσυζήτηση, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτήν. Χρειαζόμαστε αξιολόγηση, χωρίς αξιολόγηση εγώ δεν είμαι πρόθυμη να κάνω οτιδήποτε και μου είναι παντελώς αδιάφορο για ποιο σύστημα PNR μιλάμε. Είτε αφορά τον Καναδά, δεν ξέρουμε ποιον συζητάμε, καθόλου δεν με νοιάζει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε Κορνίλια Σκιώδης για το Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, έχω εκνευριστεί που συμπεριλαμβάνεται αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ψηφίσαμε όχι πέρυσι. Δεν βλέπω να υπάρχουν νέα στοιχεία στην πρόταση. Για ποιο λόγο έχει συμπεριληφθεί στη διάταξη. Τι συνέβη έκτοτε. Πέραν των όσων είπε η Κορνέλια, μέχρι πριν από ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο, μόνο ένα κράτος μέλος είχε σύστημα PNR, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο χρησιμοποιούσε πλήρως. Κανένας άλλος δεν το είχε. Από τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το είπε πολύ ευγενικά η Κορνέλια, ουσιαστικά χρηματοδότησε τη δημιουργία εθνικών συστημάτων. Ε, όπως το καταλαβαίνω εγώ αυτό, ονομάζεται δωροδοκία, το να δίνεις χρήματα στα κράτη-μέλη για να δημιουργούν εθνικά συστήματα, ώστε ξαφνικά να υπάρχει μια ανάγκη εναρμόνιση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα λόγο να φτιάξουμε μια οδηγία, ονομάζεται δωροδοκία. Χρηματισμό. Εσχρό τρόπο θεωρώ για τη χάραξη πολιτικών και νόμων. πώ θα το εξηγήσω στου πολίτε. Πέραν αυτών η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι πολλά κράτη-μέλη που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση αυτή έχουν αμφισβητούμενη νομική βάση για τη συλλογή δεδομένων PNR. Παρεμπιπτόντω, ακόμα περιμένω τις πληροφορίες που έχω ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα να μάθω χώρα προς χώρα τι συμβαίνει. Δεν μου έχει στείλει κανεί αυτές τις πληροφορίες. Τώρα όσον αφορά το κατά πόσο αιτιολογείται η ύπαρξη μιας ε, οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανείς δεν σταματά τα κράτη-μέλη, μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους συστήματα, τα PNR μόνα τους ε, είναι ελεύθερα, μπορούν να ανταλλάξουν όσα δεδομένα θέλουν. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε οδηγία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν, δεν έχουμε, αν έχουμε μια οδηγία θα υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη που δεν ενδιαφέρονται να έχουν σύστημα PNR να φτιάξουν. Και να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων εδώ, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο καταψήφισε μαζικά την πρόταση του Ολλανδού Υπουργού Δικαιοσύνης για τη δημιουργία εθνικού συστήματος συλλογής PNR. Αυτό που δεν καταλαβαίνει το Ολλανδικό Κοινοβούλιο είναι ότι η συστηματική συλλογή δεδομένων PNR συμβαίνει στις κατοχώρες ούτως ή άλλες πίσω από την πλάτη τους εδώ και χρόνια. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι και θέμα επικουρικότητας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε μια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη. Και φυσικά, και εδώ επαναλαμβάνω τόσο, όσα είπαν οι προηγούμενοι, εφόσον υπάρχουν τόσα πολλά κράτη-μέλη, εν τέλει θα χρειαστεί να κάνουμε εναρμόνιση και θα χρειαστεί το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Αλλά εδώ μου φαίνεται ότι μας τη φέρνουν. Πάνε να μας παρασύρουν σε κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό. Οι αιτίε που προβάλλονται για αυτό τη δημιουργία αυτή τη οδηγία φαίνεται να είναι κινούμενο στόχο. Στη μια μιλάμε για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, στην άλλη για την καταπολέμηση τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη δημόσια υγεία, του διχαντιστέ που ταξιδεύουν προ τη Συρία. Θα ήθελα να καταλάβω γιατί μιλάμε εδώ πέρα ακριβώ. Για παράδειγμα αυτή η νέα αιτιολόγηση, τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των τζεχαντιστών που πηγαίνουν στη Συρία δεν μου φαίνεται κάτι ιδιαίτερα λογικό. Γιατί κοιτάξτε, ακόμα και το Κοινοβούλιο ψηφίσει σύντομα μια οδηγία, δεν θα έχει ακόμα υλοποιηθεί στα κράτη-μέλη, θα χρειαστεί πολύ καιρό. Να υπενθυμίσω στου συναδέλφου και σε όσου δεν ήταν εδώ τότε ειδικότερα, θυμάμαι πως μας υποχρέωσαν να υιοθετήσουμε την οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων εντός τριών μηνών. Απαράδεκτο, επειδή ήταν εξαιρετικά επίγον έπρεπε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και τους εγκληματίες. Και ξέρετε τι έγινε. Μετά από πολλά χρόνια τελικά τα κρατημέλη δεν είχαν υλοποιήσει τίποτα. Ίσως λοιπόν να μην ήταν τόσο επίγον το θέμα. Και πράγματι και εδώ συμφωνώ με τους άλλους ομιλητές. Εάν είναι τόσο επίγον το θέμα, τότε θα έλεγα στα κράτη-μέλη ανασκουμποθείτε και υιοθετήστε την οδηγία προστασία των δεδομένων. Εάν είστε ειλικρινεί για αυτή την οδηγία, αν και εγώ έχω αμφιβολίε. γιατί έχω αρχίσει να χάνω την εμπιστοσύνη μου. Ο κύριο Σίγητη, ο κύριο Κερχόπ λέει δεν είναι ρεαλιστικό, αλλά είναι θέμα πολιτική βούληση, κύριε Κερχόπ. Εάν τα κράτη-μέλη το θέλουν, μπορούν. Μπορούν μάλιστα να αποφασίσουν πάρα πολύ γρήγορα και το έχουν αποδείξει και στο παρελθόν. Αν θέλουν προστασία δεδομένων μπορούν να την αποφασίσουν αύριο, διότι το κοινοβούλιο τους έχει δώσει ήδη το μοντέλο, τίποτα δεν τα σταματά. Τώρα ένα άλλο ζήτημα εδώ. Σόφη, λέει ο Πρόεδρος, ένα τελευταίο. Ωραία. Ε, ήθελα να, να πω όσα ήθελα να πω εδώ. Τώρα, όσον αφορά την αναγκαιότητα. Μέχρι σήμερα δεν έχω δει αποδεικτικά στοιχεία για την αναγκαιότητα. Είμαι σίγουρη ότι τα δεδομένα PNR είναι χρήσιμα, αλλά δεν έχω καταλάβει για την αναγκαία. Αυτό απομένει να αποδειχτεί. Σε αντιπαραβολή με τον καθένα από τους στόχους. Είμαι πεπισμένη ότι είναι χρήσιμα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της διακίνησης ανθρώπων, αλλά αυτά τα δύο δεν είναι το θέμα, ίδιο με την τρομοκρατία και τη δημοσιογεία, απομένει να αποδειχτεί δεν έχουμε ε, δει παρά κατακαιρματισμένα αποδεικτικά στοιχεία, όχι διατραπιστικά. Και ειλικρινά έχω αρχίσει να σχηματίζω την εντύπωση ότι οι αστυνομικές αρχές ε, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Δεν υπάρχει λόγος να μην έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, απλά δεν μοιράζονται μαζί μας τις πληροφορίες. Αυτό είναι το ευρύτερο πρόβλημα. Τώρα, για να σας πω το συμπέρασμά μου, κύριε Πρόεδρε, να πω για μια φορά αυτό που πιστεύω Τέλο και αυτό είναι θέμα αρχή. Ο κύριο Κερχόπ είπε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιε ευαισθησίε. ορισμένε χώρε στο παρελθόν έδωσαν υπερβολικέ εξουσίε στις κυβερνήσεις για ελέγχους ε, των πολιτών του και εμεί δεν το κάνουμε πια. Να σα θυμίσω ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα κράτο μέλο το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά και το οποίο χρησιμοποίησε αντιτρομοκρατική νομοθεσία για να εκφοβήσει δημοσιογράφους το γνωρίζουμε ποιος είναι, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε αυτές τις ε, τακτικές. Να είμαστε δίκαιοι προς τον Αξέλ θα πρέπει και εκείνος να έχει τον ίδιο χρόνο όπως και οι άλλοι σκιοδησηγητές. Προσοχή όμως, οι άλλοι ομιλητές θα έχουν ακόμα λιγότερο χρόνο γιατί έχουν προνομιακή μεταχείριση οι σκιοδησηγητές και τελικά να έχουμε και στο τέλος αρκετό χρόνο για να επανέλθουμε. Δεν φαίνεται το τέλος πρόκειται για πρώτο γύρο συζητήσεων για το θέμα. Οπότε να έχετε υπομονή συνάδελφε. Άξελ, και εσύ τώρα έχεις χρόνο τον ίδιο όπως και οι άλλοι σκιοδοσηγητές. Άξελ, σας ευχαριστώ. Η εργασία των υπηρεσιών εφαρμογή του νόμου παρεμποδίζεται εφόσον δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να αναλύουν τα δεδομένα. Σήμερα λοιπόν αυτό που είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του νόμου είναι να χρησιμοποιεί κανείς στοιχεία που προκύπτουν από αναλύσεις και δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ε, εγκληματίες να φεύγουν ανόχλητοι το ποινικό δίκαιο και η εφαρμογή του νόμου σήμερα έχουν φτάσει στα λειτουργικά τους όρια. Το επαναλαμβάνω. Στο ποινικό δίκαιο και στον τομέα εφαρμογής του νόμου έχουμε φτάσει στα λειτουργικά μας όρια. Άρα δηλαδή σχεδόν σε κάποιους τομείς ε, δεν θα μπορούμε να εφαρμόζουμε τον νόμο ως κράτος, διότι δεν έχουμε πια στη διάθεσή μας δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν κατά την άποψή μου ως νομοθέτες καλούμεθα να διαφυλάξουμε αυτή την ισορροπία, δηλαδή την χρήση σημαντικών δεδομένων που έχουν σημασία για την προστασία των πολιτών. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η οργανωμένη εγκληματικότητα, η τρομοκρατία, ε, ο εξτρεμισμός προς αριστερά ή προς δεξιά που εκρήγνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμείς τι κάνουμε, συζητάμε για την αναλογικότητα. Οι εχθροί του συστήματος εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τελικά αυτό που πρέπει να πούμε είναι υπάρχουν δύο πράγματα. Είτε είναι κανείς κατά της διατήρησης ε, των δεδομένων και να ξέρετε θα προχωρήσει το ποινικό δίκαιο είτε από την άλλη που είναι πιο λογικό θα επιτρέψουμε τη χρήση των δεδομένων και μετά θα υπάρχουν τα απαραίτητα όργανα ελέγχου ή διασφαλίσεις για να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα των πολιτών για να μπορούμε αν θέλετε και να αποφύγουμε την κατάχρηση. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε βεβαίως και να διαφυλάσσουμε και την αναλογικότητα. Μπορεί να υπάρχει ένα ε, ειδικό δικαστικό όργανο, ε, μπορεί να υπάρχει κάποια διαγραφή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά θα μπορούμε να τα επηράσουμε και παρόλα αυτά θα κατορθώσουμε να προχωρήσουμε. Και για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν γενικά αποθηκευμένα στοιχεία. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, τότε κατ' ουσίαν εγκαταλείπουμε το μονοπόλιο του κράτους σε αυτό το τομέα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν απέκλεισε το να μην μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αποθηκευμένα στοιχεία. Λέει μόνο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά εφόσον υπάρχουν και απαραίτητες διασφαλίσεις. Και αυτό είναι πολύ λογικό. Και το είδαμε από τα παραδείγματα, τα εύγλωτα, από τη Μεγάλη Ιταλία και τις ΗΠΑ, ότι ας πούμε στον αεροπορικό τομέα εκεί σημειώθηκε επιτυχία. Και χρειάζεται κανείς αυτά τα δεδομένα, γιατί βοηθούν στην ανάλυση. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο αυτά τα δεδομένα να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο και δεν πρέπει εκ των προτέρων να τα αποκλείουμε όλα αυτά, απλά να έχουμε λογικές διασφαλίσεις. Όπως όμως σε επίπεδο αρχής γενικά λέει όχι, αυτός θέτει σε κίνδυνο το να μην υπάρξει κανένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν μόνα τους γιατί, γιατί εμείς δεν θα είμαστε σε θέση να έχουμε ευρωπαϊκό κανονισμό. Και μάλιστα για να γίνουν αυτά τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούνται. Η προστασία λοιπόν των δεδομένων, ο κανονισμός αυτός δεν αποτελεί προϋπόθεση γιατί η προστασία των δεδομένων ρυθμίζει την χρήση δεδομένων ε, με συγκεκριμένα άτομα, όχι όμως γενικά για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε, δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει να επιτρέψουμε την χρήση των δεδομένων γιατί δεν απαγορεύεται να γίνεται κάτι τέτοιο από τα κράτη-μέλη. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει ένα νέο σύστημα. Αν δεν υπάρχει είναι κακό για τους πολίτες, κακό για την διεθνή εγκληματικότητα, δηλαδή το να κοιτάμε συνεχώς την αναλογικότητα χωρίς ε, να λαμβάνουμε και τα απαραίτητα μέτρα. Okay, thank you, Axel. Ευχαριστούμε, Άξελ. Λοιπόν, συναδέλφοι, αντιμετωπίζω ένα προβληματάκι. Ήθελα ο συνάδελφος ο κ. Κερκόπ να επανέλθει και για τις ερωτήσεις ε, και για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά έχουμε στις 3 Δεκεμβρίου μια παρουσίαση από τον Επίτροπο τον κ. Αβραμόπουλο όπου θα παρουσιάσει τους λόγους για τους οποίους συζητάμε αυτό το θέμα και το έχουμε συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη. Αλλά έχω ένα προβληματάκι, πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 12.30. Απομένουν ελάχιστα λεπτά για τη διερμηνία, αλλά έχω στον καταλογό έξι ομιλητέ. Να ρωτήσω αν κάποιος από του συναδέλφου θα έχει την ευγένεια να με βοηθήσει και να παραιτηθεί του χρόνου μιλιά στο Άννα. Ευχαριστώ, Κάρλος ευχαριστώ. Κάποιο άλλο, δεδομένου ότι οι σκιώδει έχουν μιλήσει για εσά. Κάποιο άλλο θα ήθελε να παραιτηθεί του χρόνου του. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Τόμαζη. Κύριο Μπέκερ, ναι, ευχαριστώ. 30 δευτερόλεπτα. Η ασφάλεια είναι πολύ σημαντική, δεν μπορούμε να την αγνοούμε. Πρέπει να την προσεχούμε, αλλά σεβόμενοι τον νόμο. Όσον αφορά τα PNR, πρέπει να φροντίσουμε να μην πέσουν τα, οι σε λάθος χέρια με το σύστημα PNR. Εφόσον λειτουργεί σωστά, θα βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τη διακίνηση ναρκωτικών και ανηλίκων και θα δυσκολέψει τις μεταβάσεις ανηλίκων στη Συρία όπως είχαμε πρόσφατα. Τερέζα, 30 δευτερόλεπτα. Τερέζα, εκτός μικροφώνου. Κύριε Ντίας Δεμέρα, εσείς έχετε το λόγο. Ο κύριος Ντίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να δούμε αν θα μπορούσα να σας ε, βοηθήσω για με αυτό το τελευταίο σχόλιο. Ε, μίλησαμε υπέρ, μίλησαμε και κατά και εγώ θα ήθελα να εισφέρω μια ιδέα μου σε σχέση με το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Δεν σας κρύβω ότι συμφωνώ με το PNR, το ευρωπαϊκό. Ε, θεωρώ ότι είναι κάτι το πετυχημένο. Για να δούμε όμως τι γίνεται. Έχουμε δεδομένη την απόφαση της 8 η Απριλίου θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Επίσης έχουμε δεδομένη την ψηφοφορία της Επιτροπής της 25ης Απριλίου μετά την απόφαση. Οπότε και έχουμε το 30, 25, 5, δηλαδή 30-30 είναι η ψήφος των πρασίνων. Για να δούμε όμως. Τι θα κάνουμε τώρα. Κάτι γνώμη μου ε, σύμφωνα με το δίκαιο έχουμε τις εξής εναλλακτικές ε, στο πλαίσιο της ίδιας νομοθετικής πρότασης ο εισηγητής, ο κύριος Κερκόπ θα παρουσιάσει την πρότασή του ως εισηγητής και, ε, και αν θέλει θα κάνει κάποια τροποποίηση λαμβάνοντας υπόψη κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου του Απριλίου και κατόπιν θα ανοίξει προθεσμία με τις τροπολογίες ώστε να μπορούν οι βουλευτές να ακολουθήσουν την συνήθη διαδικασία. Δεύτερη εναλλακτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τώρα διασκέπτεται έτσι κάνει πάντα. Τα σκέφτεται καλά όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει λοιπόν να κάνει κάποια τροποποίηση στην πρόταση της πριν δε εμείς θα πρέπει να περιμένουμε άρα να έρθει η πρόταση καινούργια και κατόπιν ο κύριος Κέρχοπ κατόπιν θα λάβει υπόψη την πρόταση και θα ακολουθήσουμε την συνήθεια διαδικασία. Άρα, ε, τι γίνεται τώρα. Ο κύριος Κέρχαπ ε, ταχαίως τις αμέσως μέρες θα πρέπει να μιλήσει με τους κοιόδες ηγητές. Να διαπιστώσει ο κύριος Κέρχοπ ε, τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Για να δούμε το χρονοδιάγραμμα κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τη σημερινή συζήτηση. Έχουμε την, την, την συνάντηση του Κέρχο με τους, ε, με τους σκιώδες. Στις 3 θα έρθει ο Επίτροπος, ο κύριος ε, Αβραμόπουλος, ε, το μεσημέρι για να μας πει ακριβώς ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την δικαστική απόφαση της 8ης 3 και 4 Δεκεμβρίου επίσης πρόκειται εδώ να έχουμε τον ε, Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών και ή τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών ούτω ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον ε, αντίκτυπο της συνέπειας ενός ευρωπαϊκού PNR και επίσης για τον κίνδυνο των ε, πολεμιστών αυτών. Δε στις 11 Δεκεμβρίου η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου πρέπει να παρουσιάσουν τη γνωμοδότησή τους σε σχέση με το τι γίνεται με την απόφαση της 8ης Δετάρτου σε σχέση με την οδηγία. Άρα, τι πρέπει να γίνει, τι έχουμε, θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε τι γίνεται, 25-30 ή 30-30, όπως ήταν τότε η ψηφορία, να πρέπει να τα σταθμίσουμε. Και τι έχουμε επίσης, έχουμε αυτή την απόφαση, δεν μπορούμε να την παρακάμψουμε, θα πρέπει να την λάβουμε υπόψη αυτή την ε, απόφαση. Άρα είναι σαφές το τι έχουμε μπροστά μας. Και εσείς θα πρέπει να κρατήσετε το πιδάλιο κύριε Πρόεδρε για αυτή την ε, διαδρομή. Ευχαριστώ κύριε Διασμερά. Ευχαριστούμε που περιορίσατε τα σχολεία σας διαδικαστικά. Τίμωθη, θα επανέλθω σε εσάς τώρα. Είναι δύσκολο το καθήκον σας. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε σε όλα τα σχόλια των σχεδόν. Τερέζα, θα παραιτηθείτε του χρόνου σας. να σας ζητήσω να παρεκθείτε του χρόνου σας. Δεν έχουμε χρόνο, ρωτάει η κυρία Χιμένας. Όχι, δεν πειράζει. Αν είναι απαραίτητο, δεν θέλω να πάρω το χρόνο του Τιμωθή. Αν δεν σας πειράζει, λέει ο πρόεδρος μια άλλη φορά, να επανέλθουμε στον Τιμωθή γιατί έχουμε λίγα λεπτά. Αν δεν ε, έχουν πρόβλημα οι να υπορβούν λίγα λεπτά το χρόνο τους, θα τους είμαστε ευγνώμονες. Τίμωθη, παρακαλώ ειλικρινά κύριε Πρόεδρε με το χρόνο που έχουμε εδώ και δεν θέλω να κρατήσω τις ερμηνείς εδώ. Έχουμε ελάχιστο χρόνο τώρα για τον εισηγητή. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα τα ζητήματα. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω ούτως ή άλλως με τους κοιόδης για ορισμένα από τα ερωτήματα που έθεσαν, έθεσαν σήμερα το πρωί για να δω κατά πόσο μπορούμε να τα συζητήσουμε απευθείας. Ήθελα απλά να επισημάνω δύο πράγματα, αν μου το επιτρέπετε. Κάποια από αυτά τα πράγματα είναι νέο υλικό και άλλα είναι παλιό. Πρέπει να πω ότι, ξέρετε, ο κόσμο προχωράει. Τα πράγματα σήμερα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν από ένα-ενάμιση χρόνο. Οι απειλέ είναι πολύ διαφορετικέ. Και να απαντήσω στη Σοφή λέγοντα ότι όποιο έχει έρθει εδώ επαγγελματία του τομέα και γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει με τα εγκλήματα και του κινδύνου, έχει ξεκαθαρίσει ότι μία συμφωνία PNR ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμεύει ιδιαίτερα για τις αστυνομικέ αρχές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι νομοθέτης, εκπροσωπώ μια χώρα συγκεκριμένη, αλλά ταυτόχρονα αυτό για το οποίο μιλάμε εδώ δεν αφορά ε, εθνικούς εγωισμούς. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον όλων των πολιτών της Ευρώπης. Και μου φαίνεται υποκρισία, και δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, θεωρώ υποκρισία να χρησιμοποιείται διατήρηση των δομένων για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ε, παιδιών. Έχουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα εδώ, αν όχι υψηλότερα από αυτά που προτιθέμεθα να υιοθετήσουμε στις διαπραγματεύσεις μας για τον νέο κανονισμό Ευρωπόλ για την τέταρτη οδηγία για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κανείς δεν μου αντιτέθηκε τόσο πολύ σε εκείνη την πρόταση όπου ουσιαστικά ζητάμε περισσότερες πληροφορίες από τους ανθρώπους ιδιωτικής φύσης. Το οποίο θα έπρεπε να μας ανησυχεί στην οδηγία για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Κανείς δεν κάνει αυτές τις ερωτήσεις εκεί, τις κάνει εδώ. Και πρέπει κανείς να αναρωτηθεί γιατί. Γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ας κάνουμε ό,τι κάνουμε για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και με τις δικές μου προτάσεις για να είμαστε λογικοί και να μην ε, υποπίπτουμε σε υποκρισία. Είναι εκνευριστικό. Εγώ υπήρξα ξεκάθαρος με όλους, έκανα τεράστιες προσπάθειες για να βρω τι πρότυπα ασφαλείας έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας ώστε να γνωρίζουμε ότι όταν ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση της προστασίας των δεδομένων οι διασφαλίσεις αυτές φυσικά και οι διατάξεις θα συμπεριληφθούν και σε αυτή την οδηγία. Τίποτα παραπάνω. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε σας είμαι ευγνώμων για τις παρατηρήσεις σας για το μέλλον, για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στο μέλλον, το λαμβάνω υπόψη, αλλά στο μεταξύ κύριε Πρόεδρε πιστεύω ακράδαντα ότι είναι σημαντικό. Εγώ ασχολούμαι με αυτό το φάκελο εδώ και δυόμιση χρόνια και τη Σόφη δεν της αρέσει. Πολλά πράγματα τη Σόφη υπήρξαν στην ημερήσια διάταξη. Εγώ πήρα ένα πράγμα σε αυτή την καταραμένη ημερήσια διάταξη, αν μου το επιτρέπετε να το πω. Ένα θέμα, με ένα θέμα ασχολήθηκα σε αυτή την ημερήσια διάταξη και είμαι πεπισμένο για την αξία του. Ξέρω ότι πρέπει να πείσω και άλλου, ίσω να μην έπεισα ποτέ τη σόφη, αλλά τώρα δεν μπορεί να αμφισβητεί το δικαίωμά μου να συμπεριλαμβάνομαι σε αυτή την ημερήσια διάταξη, αν δούμε τι συμπεριλαμβάνει αυτή στην ημερήσια διάταξη. Ορισμένα τα οποία μάλιστα δυσκολεύομαι να καταλάβω. Λοιπόν, η αλήθεια είναι τώρα δεν θα επιμείνω άλλο. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Θα προσπαθήσω να παράσχω τύπωση που να ικανοποιεί όλου όσου μίλησαν σήμερα το πρωί και σα ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσετε σήμερα. Ευχαριστούμε να εξηγήσω στου συναδέλφου ότι η λέξη καταραμένο, flipping, είναι μια εξαιρετική ε, λέξη στα αγγλικά, η λέξη flipping που ανέφερε ο κύριο Συγητή. Απολύτω δεκτή. Και να πω στα νέα μέλη ότι το PNR είναι ένας από τους πιο αντιφατικούς φακέλους που έχουμε. Καλό είναι λοιπόν να συζητηθεί από τους συντονιστές και για τα διάφορα σημεία που ανέφεραν οι συναδέλφοι για το μέλλον. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα. Είναι καλύτερο να ασχοληθούν με αυτό οι συντονιστές, με τους κοιόδης και τον εισηγητή. Πιστεύω ήταν επικοδομητικό που είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων ώστε να επαναφέρουμε το ζήτημα στις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής. Ευχαριστώ όλους σας. Καλό μεσημέρι.